Okay, Φίλοι μου, καλώς επιστρέψατε στις Βρυξέλλες. Να ξεκινήσουμε με την έγκριση της εμερήσιας διάταξης, η οποία εγκρίνεται χωρίς αλλαγές. Ωραία. Προχωρούμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις της Προέδρου. Η διερμηνία σήμερα προσφέρεται σε όλες τις γλώσσες εκτός των μαλτέζικων, βουλγαρικών και κροατικών. Τα βουλγαρικά θα υπάρχουν στην συνεδρίαση της Τετάρτης το μεσημέρι με την παρουσία του Βουλγαρου Υπουργού. Επισκέπτες ε, θα υπάρξουν 21 επισκέπτες ασκούμενοι στη μετάφραση της Digitrad στο Λουξεμβούργο και θα παραστούν στη συνεδρίαση της Τετάρτης έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 27-28 Νοεμβρίου. Δεν, δεν έχει κανείς κάποια προσθήκη να ζητήσει από ό,τι βλέπω. Οπότε περνάμε στο σημείο 4 της ημερησίας. Ενημέρωση για, τους τρέχοντες, για τις τρέχουσες διαθεσμικές διαπραγματεύσεις. Για την απόσπαση των εργαζομένων είχαμε ενημερωθεί και την τελευταία φορά τίποτε άλλο να προσθέσουμε σήμερα. Απλώς να γνωρίζετε ότι απόψε θα έχουμε τριμερή και θα είναι ο πέμπτος γύρος. Μετά από αυτά φτάνουμε στο σημείο 5 στην ημερησία για την προστασία των εργαζομένων και τους κινδύνους από τα καρκινογόνα και τα μεταξαλιογόνα στο, στο χώρο εργασίας. Ελπίζω να ακούσατε τι είπα. Ε, να δώσω λοιπόν το λόγο στον εισηγητή μας τον κύριο Ρολά. Ευχαριστώ Πρόεδρε πράγματι. Πρόκειται για το δεύτερο τμήμα της αναθεώρησης της οδηγίας για την προστασία των εργαζομένων από τα καρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τις τροπολογίες που υπέβαλαν. Κάτι λιγότερο από 120 τροπολογίες, οι οποίες είναι τροπολογίες ποιοτικές Βασιστήκαμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν ενδιαφέρουσα σε κάθε περίπτωση και Ήδη το έχω πει, αλλά το επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω. Είναι σημαντικό η Επιτροπή και η Επίτροπος Τάισεν να συνεχίσουν αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να πάψουν να προστατεύουν τους μισθωτούς εργαζομένους από τα καρκινογόνα και μεταλλαξιογόνα. Εδώ και 10 χρόνια αλλαγή δεν υπήρξε στην ισχύουσα νομοθεσία, οπότε είναι σημαντικό να προχωρήσουμε. Υπάρχει μια δυναμική πια τάση και το λέω γιατί βλέπουμε κάτι που προχωράει στο χρόνο. Είχαμε ένα πρώτο τμήμα των προτάσεων, τώρα έχουμε ένα δεύτερο τμήμα που έχει προεξαγγελθεί και διαμορφώνεται μια μελλοντική θεώρηση για αυτού του είδους τους παράγοντες κινδύνου. Η αναθεώρηση όπως είχα εξηγήσει ήδη όταν το συζητήσαμε για το πρώτο τμήμα η δική μου προσέγγιση θα είναι να βασιστώ σε επιστημονικά στοιχεία, αλλά κυρίως και πρωτίστως να βασιστώ στην άποψη των ενδιαφερομένων, των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αυτοί που γνωρίζουν καλύτερα και τις απειλές κατά της υγείας και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο επιχειρήσεων, εταιριών και παραγωγικών τομέων και κλάδων. Όπως κάναμε και για το πρώτο τμήμα της πρότασης, θέλουμε να συνδυάσουμε την ε, υψηλή μας φιλοδοξία για την προστασία των μισθωτών εργαζομένων, αλλά ταυτόχρονα να παραμείνουμε και πραγματιστές ώστε να προτείνουμε εφικτές λύσεις στους διάφορους κλάδους και στις διάφορες εταιρείες. Διότι σημαντικό είναι να θεσπιστούν συστήματα που να μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και να εφαρμοστούν όντω. Για τις διάφορες τροπολογίες που έχω λάβει, πέραν της ποιότητας υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία τίνουν ε, στην ίδια Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε καλή δουλειά με βάση αυτές τις τροπολογίες και σίγουρα κάποιοι θέλουν να πάμε πιο μακριά, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στη διατύπωση, άλλοι το αντίθετο, αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να βρούμε το σωστό σημείο ισορροπίας. Το πλέον ε, σημαντικό σημείο που θα χρειαστεί να συζητήσουμε είναι το θέμα των εκπομπών των ε, εξατμίσεων δίζελ εδώ σε σχέση με τις διάφορες τροπολογίες που έλαβα μπορώ να πω ότι όλοι συμφωνούν ότι πρόκειται για ένα προβληματισμό σημαντικό. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις στις απόψεις των συναδέλφων, δεν έχουν όλοι την ίδια θεώρηση αλλά το θέμα είναι πώς όλον αυτόν τον προβληματισμό θα τον αξιοποιήσουμε. Διότι κάποιοι θέλουν όρια και τιμές έκθεσης πολύ δεσμευτικούς και αυστηρούς, άλλοι πιστεύουν ότι μπορούμε να συνεχίσουμε την έρευνα και τη μελέτη για το θέμα και όσο το δυνατόν συντομότερα να εφαρμόσουμε όρια που να είναι δεσμευτικά. Κάποιοι άλλοι, όπως και εγώ ίδιος, προτείνουν να δουλέψουμε με βάση την αξιολόγηση για, τα βασικά, ε, για τους βασικούς για τους στοιχειακούς άνθρακες και εδώ θα κάνουμε την πιο πολλή δουλειά. Πάντως, νομίζω ότι οι προθέσεις ε, όλων των συναδέλφων, ακόμη και αν έχουν διαφορετικές ιδέες για το τι λύση θα βρούμε, περίπου συγκλίνουν. Αυτό που σε κάθε περίπτωση μου φαίνεται σημαντικό σε αυτή τη δουλειά και γι' αυτό το ανέφερα και προηγουμένω, την δυναμική τάση αυτή, είναι ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το, τη συνέχεια στο χρόνο που έχει υπάρξει με την πρόταση αυτή. Δηλαδή, στο δεύτερο τμήμα δεν ξεκινάμε από το μηδέν, μπορούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που έχει αρχίσει. Δεν χρειάζεται να φορτώσουμε όλα τα φορτία στο ίδιο αγώγι, αν μπορώ να το πω έτσι, ε, γιατί μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δουλειά που έχει προηγηθεί. Και θα μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε και στο μέλλον. Για τις τροπολογίες λοιπόν αυτές νομίζω μπορούμε ήδη να συζητήσουμε από αυτή την εβδομάδα για να προοδεύσουμε εντάχει και γιατί έχει προαναγγελθεί και το τρίτο τμήμα της νομοθεσίας. Θέλουμε λοιπόν η δυναμική αυτή τάση, ταχύτητα να συνεχιστεί και να μην τη φρενάρουμε όπως έγινε και με το πρώτο τμήμα. Και το τελευταίο που θέλω να πω εν είδη είναι ότι έχω την πεποίθηση και με τη Μαρίτα το γνωρίζω, θα εργαστούμε πολύ καλά και θα έχουμε πλήρη και ικανοποιητικά αποτελέσματα και το ίδιο και στο επίπεδο του τριμερούς διαλόγου. Θα είμαστε περίπου οι ίδιοι στην ομάδα που θα διαπραγματευτεί στον τριμερή διάλογο, οπότε νομίζω θα εκφράσουμε το ίδιο θετικό πνεύμα συνεργασίας ως τώρα, που εκφράσαμε ως τώρα. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ρολά. Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για το έργο σας ε, σε ό,τι το σχέδιο έκθεσης που είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας και συζήτησης. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κομισιόν για τις προτάσεις της ε, που θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε από κοινού. Όπως μπορείτε και εσείς να δείτε από τις δικές μου τροπολογίες, ε, τις τροπολογίες που κατέθεσα ως και συγγήτρια, στηρίζω τις προτάσεις του κυρίου Ρολά σε ό,τι αφορά τους ε, πολυκυκλικούς ε, αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Ε, από ό,τι κατάλαβα το ίδιο κάνει και το Συμβούλιο και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης για να βελτιωθεί η οδηγία. Εν γέννη θεωρώ ότι η διαδικασία που ακολουθεί η Κομισιό θα πρέπει να γίνει σεβαστή, εκτός αν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να μην γίνει αυτό. Άρα πρώτα θα πρέπει να δούμε τα επιστημονικά στοιχεία μέσω της ε, Επιστημονικής Επιτροπής για τα Όρια Επαγγελματικής Έκθεσης της ΚΟΕΛ και μετά τους κοινωνικούς εταίρους. Έτσι έχουμε μια πολύ ισχυρή, στέρη βάση εργασίας και έτσι έχουμε εργαστεί και μέχρι τώρα. Ταυτόχρονα, σίγουρα όλες οι προτάσεις έχουν και πολιτικό χαρακτήρα που σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε εντελεχώς και να εμπαθύνουμε σε αυτές τις προτεραιότητες. Από τη δική μου οπτική γωνία, όταν η επιστημονική κοινότητα ή οι κοινωνικοί εταίροι μας στείλουν ε, χειρά μηνύματα ότι τα όρια θα πρέπει να είναι είτε πιο ε, αυστηρά είτε λιγότερο, θα πρέπει να τους ακούσουμε και θα πρέπει βέβαια μετά τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις με αυτούς να καταλήξουμε στις δικές μας αποφάσεις. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι και ε, το πνεύμα που διέπηκε τον κύριο Ρολά και εγώ θεωρώ ότι έτσι πρέπει να προχωρήσουμε στη σημαντική αυτή έκθεση. Και άλλωστε αυτός είναι και ο λόγος ακριβώς ε, που Πιστεύω ότι για το ντίζελ, τα καυσαέρια δηλαδή, κινητήρων ντίζελ, πρέπει να μπει οριακή τιμή έκθεση και προτείνω στη δίκτυ να χρησιμοποιηθεί ω τυχιακό άνθρακα. Προτείνω επίση και το διοξίδιο του αζότου να είναι ένα δείκτη ε, για να καλύπτει και τις σχετικούς ε, κινητήρες. Ε, αυτό το λέει και η έρευνα που έχει γίνει από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων των σκανδιναβικών χωρών για την αξιολόγηση κινδύνων από τα κασέρια και επίσης η Επιτροπή Ολλανδική για την Επαγγελματική Ασφάλεια. Υπάρχει επίση ενημέρωση για αυτά που λέει η ΣΚΟΕΛ, η Επιστημονική Επιτροπή για τώρα Επαγγελματική Έκθεση, ό,τι αφορά ε, τη, τα καυσαέρια κινητήρων δίζελ. Περιμένουμε να δημοσιοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία. Ούτω ή άλλω, από το 2012, η Παγκόσμια Οργάνωση Υγεία ξεκάθαρα έχει επισημάνει ότι από τα καυσαέρια αυτά προκαλείται καρκίνο. Πάνω από 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι στον κόσμο είναι εκτεθειμένοι σε αυτά τα καυσαέρια. Υπάρχει επιστημονική βάση και μάλιστα υπάρχουν οριακέ τιμέ ε, για τα καυσαέρια από κινητήρε δίζελ σε ορισμένε χώρες, μέλη. Γι' αυτό και εγώ υποστηρίζω στεναρά την άποψη του κυρίου Ρολά και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε ένα βήμα προς την ε, καλύτερη προστασία των εργαζομένων. Και έχουμε την ευκαιρία με αυτή την έκθεση. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον επόμενο σκιώδη, συγκεκριμένα στην κυρία Μακιντάρη, η οποία εκπροσωπεί την ομάδα ECR, τους Ευρωπαίους Συντηρητικού. Έχετε το λόγο. Κύριε Μακιντάρ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας, τον κύριο Ρολά. Πρόκειται για τη συνέχεια μιας διαδικασίας ε, που πιστεύω όσο συνεχίζεται και εμείς θα βελτιωνόμαστε. Σίγουρα οι ωριακές τιμές της πρότασης της Κομισιόν είναι αποτέλεσμα πολλών ετών αναλυτικής δουλειάς, αξιολόγησης ε, και check-up, αν μπορώ να τα πω έτσι, fitness checks. Και πιστεύω ότι η διαδικασία για τον καθορισμό των ωριακών τιμών ε, είναι αρκετά σοβαρή και πρέπει να την υποστηρίξουμε. Γιατί ο στόχος μας είναι να βασιζόμαστε σε στοιχεία, να τα βλέπουμε αναλογικά τα πράγματα, οι οριακές τιμές να είναι μετρήσιμες και να είναι και εφικτές πιστεύω ότι η ανάληψη δράσης για μείωση του αριθμού θανάτων και άλλων προβλημάτων υγείας λόγω της έκθεσης ε, σε επικίνδυνους παράγοντες, ε, μεταλλαξιογόνους ε, ή καρκινογόνους είναι κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και το ρόλο των καλών πρακτικών, όπως αυτές που βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, με τη Συμφωνία Κοινωνικού Διαλόγου, που ε, μιλάει για την εφαρμογή της οδηγίας περί μεταλλαξιογόνων και καρκινογών παραγόντων. Έχω καταθέσει τις τροπολογίες 43-119 ακριβώς σε αυτό το πνεύμα. Νομίζω ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε θα πρέπει να έχουν ως στόχο τον έλεγχο και τη διατήρηση των ε, εκθέσεων σε όσο το πιο χαμηλά επίπεδα. Άρα, ορικές τιμές έκθεσης θα πρέπει να οριστούν σε επίπεδο που θα βοηθούν τη διαχείριση των κινδύνων από την έκθεση έκθεση σε δυνητικά επικίνδυνε ουσίε. και νομίζω ότι ο τελικό μα στόχο θα πρέπει πάντοτε να είναι τα κατώτατα δυνατά επίπεδα έκθεση κατώτερα και από αυτά τα οποία προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει ενεργά να επενδύουν στην επιστήμη, να ενθαρρύνουν τι επιχειρήσει να προσπαθούν να επιδιώκουν πάντοτε το χαμηλότερο δυνατό επίπεδο έκθεση. Και πιστεύω ότι και εμεί δεν θα πρέπει αυθαίρετα να ορίζουμε οριακές τιμές τόσο χαμηλές, που τελικά αυτές να μην μπορούν ούτε να μετρηθούν αλλά ούτε και να επιβληθούν, να εφαρμοστούν. Θέλω λοιπόν να τονίσω και μια άλλη τροπολογία που έχω καταθέσει, την υπαριθμόν 28 αλλά και την τροπολογία μου παριθμό 42 και τις τροπολογίες 22, 30, 34 και 41 θα τις υποστηρίξω. Οποιαδήποτε νέα πρόταση η αλλαγή των οριακών τιμών θα πρέπει να υποβληθεί στην ίδια αυστηρή διαδικασία αξιολόγηση με αυτή που ίσχυσε τον αρχικό καθορισμό αυτών των οριακών τιμών και για την πρόσθεση ουσιών. Πιστεύω ότι το ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείτε. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η ομάδα μας έχει κάποιες ανησυχίες με την πρόταση του εισηγητή και με κάποιες από τις κατατεθείς τροπολογίες για την εισαγωγή ορίων έκθεσης, επαγγελματική έκθεσης σε ό,τι αφορά τη, τα καυσαέρια κινητήρων diesel. Πολλές είναι, αλλά 8, 20, 21, 51, 52, 55, 93... 114, 115, 116 αυτές είναι σημαντικότερες. Υπάρχουν πολλές σχετικές τροπολογίες. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην προχωρήσει στη συμπερίληψη αυτών ε, των καυσαερίων για λόγους που τους λέει στο 4-2-3 τμήμα της μελέτης αντικτύπου που συνοδεύει την πρότασή της. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτούμε πολύ προσεκτικά για το κατά πόσο θέλουμε να πιέσουμε να περάσουν αυτές οι τροπολογίες στη δεύτερη φάση. Επιπλέον, η ΣΚΟΕΛ, η Επιστημονική Επιτροπή για το ώρα επαγγελματική έκθεση, πάντα λέει ότι το να έχουμε ένα κατόφλι για, τις, ε, για την έκθεση των εργαζομένων στα κασέρια αυτά δεν είναι εφικτό αυτή τη στιγμή. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε όμως μια λύση. Ίσως στη θέση του Κοινοβουλίου θα έπρεπε να συμπεριληφθεί η απέτηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τα πράγματα το έχουμε κάνει και για τα θέματα αναπαραγωγικής υγείας που δίνουμε τη δυνατότητα έτσι στην Κομισιόν να επανέλθει. Άρα η τροπολογία 53 η δική μου νομίζω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και θα στήριζα και την 50, 84 και 86 τροπολογίες άλλων συναδέλφων. Ένα άλλο επίμαχο, αμφιλεγόμενο θέμα κατά εμάς είναι η πολυκυκλική αρωματική υδρογονάνθρακης. υπάρχει σκέψη να επεκταθεί ε, το εύρος αυτής της ε, νομοθεσίας και να έχουμε κάποιο σωρικές στιγμές και για αυτούς τους ναι. υδρογονάνθρακες. Ναι, μεν υπάρχουν ανησυχίες για το πώς επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων, αλλά εγώ νομίζω ότι απαιτείται να έχουμε πρώτα στη θέσή μας περισσότερα στοιχεία και μετά να δούμε κατά πόσον πρέπει να επεκτάθει το πεδίο εφαρμογή και να καλύψει και αυτέ αυτές τις Γι' αυτό στηρίζω την τροπολογία 9 του εισηγητή, καθώς και τι τροπολογίε 59 και 87 που λένε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει, να προβεί σε περισσότερο έργο επ' αυτού. Επίσης θεωρούμε ότι η αναλογικότητα, το εφικτόν, η σκοπιμότητα είναι στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να έχουμε αποτελεσματικέ ορικέ τιμέ που μπορεί να είναι και εφικτέ. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και θα ανταλλάξουμε φαντάζομαι περισσότερες λεπτομέρειες και στι συνεδρίαση που θα έχουμε μεταξύ των σχεδόν αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Ευχαριστώ, Ανθέα. Καλβέτ Σαμπον. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα γαλλικά θα συγχαρώ απλώς τον εισηγητή για την εξαιρετική του δουλειά και την πλατφόρμα που δημιούργησε, γιατί θα είναι πολύ πιο εύκολο έτσι να καταλήξουμε σε συμφωνία. Αξιοπερίεργο από τον κύριο Ρολά, αλλά αυτή τη φορά έπιασε και θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου, φίλε μου. Διευκολύνεις πολύ τη δουλειά μας. Τώρα θα περάσω στα ισπανικά για να πω ε, κάποιες παρατηρήσεις μου. Γιατί έχω υποβάλλει τροπολογίες από την πλευρά των φιλελευθερών. Ισπανικά λοιπόν τώρα. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει αυτός ο φάκελος για την υγεία των εργαζομένων. Δηλαδή, οριακέ τιμέ που καθορίζουμε κτλ. κτλ δεν θα είναι περιβαλλοντικές οριακές τιμές για την υγεία των πολιτών, αλλά για την υγεία των εργαζομένων συγκεκριμένα και θα είναι τιμέ για την έκθεση την οποία υφίστανται λόγω ε, του χώρου εργασίας τους. Άρα οι τιμές θα πρέπει να σχετίζονται πολύ περισσότερο και με το χρόνο έκθεσης. Επειδή όμως ακριβώς έχει να κάνει το θέμα άμεσα με την υγεία και όχι μόνο με το περιβάλλον, αυτό που θα θέλαμε θα είναι ε, με υπερβολική φιλοδοξία ή με εστίαση στη λεπτομέρεια να γυρίσουμε πίσω. Ε, είπατε πολύ καλά κύριε Ρολέν ότι υπάρχει μια συνέχεια γιατί έχουμε τη τρίτη φάση που έπεται. Το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι οι αξιολογήσεις, οι μελέτες αντικτύπου θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρές και σε αυτό θα επιμείνουμε, ιδίως όταν σκοπός είναι να προωθηθούν νομοθετικές αλλαγές, γιατί αυτές οι νομοθετικές αλλαγές ε, που οφείλονται σε τεχνικές πτυχές, όρια έκθεση κτλ. κτλ προκαλούν στρέβλωση μεγάλη στρέβλωση σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό ε, των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι σημαντικό. Σίγουρα πρέπει να γίνει γιατί η προτεραιότητα έχει υγεία πάντοτε, όμως ε, ε, σίγουρα κάλλιον ε, το προλαμβάνει του θεραπεύει. Και γι' αυτό θα πρέπει πάνω απ' όλα να λαμβάνουμε υπόψη σε αυτό το μεγάλο ευρωπαϊκό ιστό και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ΜΜΕ που πάντοτε θα αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες ε, στο να αντιδράσουν γρήγορα και να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ξέρουμε και ε, ότι η ανεργία και η απώλεια θέσεων εργασίας επηρεάζει αρνητικά και την υγεία των εργαζομένων. Να πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό και στον τομέα που μας απασχολεί τους καρκινόγονους παράγοντες. Επίσης, πρέπει να έχουμε πράγματι ε, στοιχεία πολύ στέρεα επιστημονικά και ή δυνατόν αυτά να είναι ομόφωνα και να μην υπάρχουν ε, αμφισβητήσεις και ενστάσεις. Γιατί τότε έχουμε μια πραγματικότητα που δεν είναι ακριβώς επιστημονική. Γι' αυτό στηρίζουμε αυτό που είπε η πρόεδρός μας. Η προεδρεύουσα καλύτερα. Δηλαδή ότι πρέπει να στηρίζονται όλα οι προτάσεις από μια αυστηρή, στέρεη επιστημονική βάση. Μετά από πολλά χρόνια αναζήτηση νομίζω ότι είναι η σωστή κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουμε. Και έρχομαι στο περιβόητο θέμα του ντίζελ. Δεν νομίζω ότι αυτό το θέμα θα έπρεπε να μας ε, εμποδίσει να καταλήξουμε σε συμφωνία, ούτε πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι ακόμη και μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, Ενίοτε δεν υπάρχει συμφωνία για το κατά πόσον ε, έχουμε το νέο ή το παλιό μοντέλο, δίζελ κτλ. Και αυτό μπορεί να μην βασίζεται κατά πάσα πιθανότητα στα επιστημονικά στοιχεία, αλλά σε συμφέροντα εντό αγωγικών. Άρα και είναι και κατανοητό. Λένε λοιπόν οι κατασκευαστέ ότι σίγουρα πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι, να υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των επιστημόνων και να μην υπάρχουν ενστάσει ή αμφισβητήσει ω προ τα στοιχεία αυτά. Και εμεί ως ε, πιθανή συμφωνία θεωρούμε ότι ε, είναι να ζητήσουμε από την Κομισιόν να συμπληρώσει τη μελέτη αντικτύπου. Να συμπληρώσει όλες αυτές τις έρευνες με απόλυτη προτεραιότητα και στον να το πιο γρήγορα. Να μην έχουμε δηλαδή μια προχειρότητα ε, με αυτό το νομοθετικό πακέτο, ε, ούτε όμως και τελικά να τα καθυστερήσουμε ε, τα μέτρα αυτά. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι ουσιαστικά ε, αυτό είναι ένα τμήμα της όλης συζήτησης που δεν θα πρέπει όμως να θέσει εμπόδια και προσκόμματα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλα αποφασιστικά με ένα λαψίχρεμα και όχι με συναισθηματισμούς, βάζοντας στο ε, προσκήνιο την υγεία των εργαζομένων χωρίς όμως να κινδυνολογούμε, αλλά να έχουμε ε, ως βάση επιστημονικά στοιχεία αποδεδειγμένα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια ακόμη φορά. Και επαναλαμβάνω την άποψή μας ότι δεν θα πρέπει αυτό το θέμα του ντίζελ να είναι επίμαχο και να αποτρέψετε την συμφωνία. Αυτό πιστεύει άλλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Καλβέ Σαμπον. Από την GUNGL δεν βλέπω τον κύριο Ρέγγι εδώ. Υπάρχει κάποιος άλλος. Τον κύριο Λέιαρίκ. Και τώρα Προχωρούμε στον επόμενο εισηγητή. Η κυρία Ντελή από τους Πρασίνους δεν είναι εδώ. Οπότε η Τζιν Λάμπερτ θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Καρή Μαντελή προεδρεύει αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Μεταφορών. Μου ζήτησε λοιπόν να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και όχι τόσο πολύ για τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Προφανώς το βασικό σημείο για μας είναι η εργασιακή έκθεση στο χώρο εργασίας των εργαζομένων για τα καρκινογόνα, με τα λαξιογόνα και τις ε, τοξικές ουσίες να ληφθεί υπόψη σε συνδυασμό και σε σύγκριση με τον γενικότερο πληθυσμό. Νομίζω ότι αυτό συνάδει με κάποια από τα σχόλια που έκαναν κάποιοι από τους συναδέλφους το απόγευμα. Επίσης, τα ευρωπαϊκά όρια έκθεσης θα πρέπει να είναι δεσμευτικά και όπως είπαν ε, οι υπόλοιποι με τις πλέον επίκαιρες επιστημονικές πληροφορίες. Άρα, ε, συστηματική αναθεώρηση χρειάζεται. Να μην ε, λάβουμε υπόψη το κατώτατο επίπεδο που μπορεί να επιτραπεί σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να είναι επιρρεπής σε health dumping, σε dumping της υγείας, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι έχουν πολύ χαμηλά πρότυπα προστασία πρέπει να γίνει αυτό και σε άλλα μέρη τη ε, εσωτερική αγορά. Επίση, χαιρόμαστε, όπω είπε και ο εισηγητή, που η συμπερίληψη του ντίζελ ε, είναι αντικείμενο συμφωνία. Τουλάχιστον αυτό θα το έχουμε. Αλλά να συζητήσουμε τι καλύτερε τιμέ ε, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ω ανώτατα όρια σε πρώτη φάση. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει σταδιακή μείωση του ντίζελ ή δυνατόν γιατί ε, ο Διεθνής Οργανισμός για την έρευνα για τον καρκίνο το έχει χαρακτηρίσει από τις πλέον καρκινογόνες ουσίες για τους ανθρώπους. Ε, έχουμε μιλήσει για μια σταδιακή μείωση μέσα σε μια πενταετία σε πρώτη φάση, οπότε θα πρέπει να ε, κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον δίζελ. Χαιρόμαστε που και άλλε ομάδε θέλουν και άλλε ουσίε να καλυφθούν από την οδηγία και ανυπομονούμε για τις συζητήσει για όλες αυτές τις ουσίε και για τις οριακέ τιμές που προτείνονται από τι διάφορε ομάδε. Για τι ε, τοξικέ ουσίε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει αρκετά για να προστατεύσει του εργαζομένου και υπάρχει καθυστέρηση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν επιλαμβάνεται εγκαίρος του θέματος. Υπάρχουν ε, εταιρείε, όπως εντυπώ στις κατοχώρες και γυναίκες που εργάζονται εκεί έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Οι ουσίες αυτές δεν καλύπτονται από την οδηγία. Θα θέλ... Μάλλον καλύπτονται από την προηγούμενη οδηγία. Θέλουμε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή, Επι... Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωση για το αν είναι ικανοποιημένοι με την ταχύτητα με την οποία όλα αυτά υλοποιούνται. Θα πρέπει να υπάρξουν επικοδομητικέ και πλήρε διαπραγματεύσει για αυτό το πολύ σημαντικό φάκελο, αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προστατεύει του εργαζομένου τη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω τη Λάουρα Αγκάρ τη πολιτική ομάδα EFDD. Μήπω την αντικαθιστά κάποιο. Όχι. Άρα, τώρα Ζωέλ Μαλάνς της ομάδας ε, Ευρώπη των Εθνών δεν είναι ούτε αυτός ή αυτή παρούσα. Άρα, επειδή έχουν τεθεί ορισμένες ερωτήσεις ευθέως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορούμε να παρακαλέσουμε τον εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Στέφαν Όλσον. Ορίστε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, καθώς και τους συζητητές και εισηγητές και τα αξιότιμα μέλη. Θα είμαι σύντομος. Άλλωστε λέχθηκαν τα περισσότερα. Υπάρχει πλήρης κατανόηση της διαδικασίας την οποία διαπιστώνω εδώ στην αίθουσά σας, άρα δεν χρειάζεται να επαναλάβω τίποτε. Είμαστε ικανοποιημένοι με το σχέδιο εκθέσεως που είδαμε, είναι καλά συνταγμένο, βασίζεται στην πολύ γερή δουλειά που έχει γίνει εδώ από την πλευρά σας για το CMD1. Τώρα, να καθησυχάσω ή πάντως να επανέλθω σε ορισμένα θέματα, διότι μιλήσατε για την recurring process. Ο ίδιος ο κ. Ρολάν το εξήγησε. Σας βεβαιώνουμε ότι πρόκειται πράγματι για μια διαδικασία που συνεχίζεται. Προχωρούμε στη μελέτη αντικτύπου που εντάσσεται μέσα στην διαδικασία αυτή. Αυτό θα γίνει τον Φεβρουάριο και ελπίζουμε η πρόταση ε, να είναι έτοιμη πριν από το Πάσχα. Προχωρούμε λοιπόν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Έχουμε διαβουλευτεί με τους κοινωνικούς εταίρους σύμφωνα και με τα άρθρα 174 και 75 της συνθήκης. Έχουμε λάβει τις απαντήσεις τους. Προχωρούμε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και τη μελλοντική τροποποίηση που θα είναι CMD4. Άρα μια διαδικασία που δεν πρόκειται να σταματήσει αλλά θα συνεχιστεί. Όπως επίσης εξήγησε ο κύριος Ρολάν, είναι μια δουλειά αρκετά δυσκίνητη. Χρειάζεται όμως να περάσουμε μέσα από τη διαδικασία της επιστημονικής επεξεργασίας, μετά διαβούλευση στην Επιστημονική Επιτροπή, Συμβουλευτική Επιτροπή, με τους ενδιαφερομένους και μετά υπάρχουν και κάποια θέματα ασφαλείας. Πρέπει να βρούμε λοιπόν μια ισορροπία και να συνεχίσουμε με τη διαδικασία αυτή. Απλώς θέλω να πω δηλαδή ότι δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε όλες τις ουσίες ταυτόχρονα Τώρα σε μια από τις τροπολογίες θα έρθει σε νέα πρόταση τη τέλη Μαρτίου. Και επίσης όπως εξηγήσατε εσείς κυρία Πρόεδρε, ακολουθούμε τη διαδικασία που προβλέπετε. Λαμβάνουμε τις επιστημονικές συμβουλές και μετά και από έλεγχο μελέτης αντικτύπου ελέγχουμε και τι έχουν συζητήσει οι κοινωνικοί εταίροι. Βέβαια τη συζήτηση την κάνετε και εσείς εδώ, με πολιτικό χαρακτήρα δηλαδή. Υπάρχει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε μαζί σας και βεβαίως και στις μελλοντικές συζητήσεις που θα διεξαγάγετε εσείς με το Συμβούλιο Υπουργών. Και μέχρι τώρα η διαδικασία για την CMD1 ήταν ε, πολύ καθαρή. Για τις για τις ρεπροτοξίνες συνεχίζουμε όπως έχει σχεδιαστεί και θα περιληφθούν στις τροπολογίες CMD1 θα υποβάλουμε δε τη σχετική μελέτη αρχές του 2019 και εκεί λοιπόν βρισκόμαστε μέσα στο χρονοδιάγραμμα να αναφερθώ πολύ σύντομα στο ζήτημα της νέψη και για ποιο λόγο εκτιμούμε τις τροπολογίες της κυρίας Μακιντάιρ. Υπάρχει μια τροπολογία που αναφέρεται στα συμβαλόμενα μέρη της Συμφωνίας έψη και θεωρεί ότι αυτά εξαιρούνται από ορισμένα μέρη της Συμφωνίας. Νομικά ωστόσο δεν νομίζω αυτό να είναι δυνατό. Δεν αρκεί δηλαδή μια τροπολογία που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Όμως η καταγραφή των συμφωνιών των κοινωνικών εταίρων και η αναβάθμισή τους νομίζω είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση γιατί εμείς υποστηρίζουμε τις συμφωνίες αυτές και ως γνωρίζετε η εφαρμογή της οδηγίας είναι αυτή που έχει τελικώ σημασία και γι' αυτό απαιτείται επιχειρήσεις και ε, εργατικές ενώσεις να συνεργάζονται. Όποια Δίποτε λοιπόν λήψη υπόψη των συμφωνιών αυτών ή των συμβάσεων αυτών ε, έχει καλο Αλλά τώρα να αναβαθμιστούμε τον τρόπο που λέτε αυτό δεν είμαι βέβαιο τι νομικά γίνεται. Τώρα ε, για του ορισμού. Αν μιλήσουμε για κοιτοτοξικά φάρμακα, πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώ για ποιο πράγμα μιλούμε. Διότι κάθε ουσία ή ορισμό που θα ενταχθεί στην οδηγία σημαίνει και άμεση αξίωση επιδότησης για τον ε, εργοδότη. Πρέπει να γνωρίζουμε λοιπόν ακριβώ για ποια πράγματα μιλούμε, να έχουμε τι επιστημονικέ ενδείξει και αποδείξει και να μπορούμε να είμαστε σαφεί. Άρα χρειάζεται κάποιο, κάποια προσοχή. Εάν εντάσσουμε νέου όρου στην οδηγία, θα χρειαστεί να γνωρίζουμε ακριβώ γιατί πρόκειται. Δηλαδή, προβλέπεται άμεση υποκατάσταση εφόσον αυτό είναι τεχνικώ δυνατό. Αυτό θα έχει βεβαίω επιπτώσει ε, στη φροντίδα προσφέρουν τα νοσοκομεία κλπ. Αν δηλαδή βάλουμε απλώς έναν όρο ή έναν αριθμό φαρμάκου μέσα στην οδηγία. Τώρα, για το καύσιμο ντίζελ νομίζω η συζήτηση σας απέδωσε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Από πλευρά κομισιών δεν θεωρήσαμε ότι υπάρχει επαρκή ασφάλεια δικαίου για να το περιλάβουμε. Ούτε υπάρχει και συμφωνία μεταξύ των ε, κοινωνικών εταίρων. Προχωρούμε λοιπόν με τη διαδικασία. Θα παρακολουθούμε και τις συζητήσεις που διεξάγετε εσείς, καθώς και τις συζητήσεις σας με το Συμβούλιο και είμαστε στη διάθεσή σας για να συνεργαστούμε μαζί σας. Ε, αρκούμε σε αυτά και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση. Thank you for that, ε, Mr. Ευχαριστώ κύριε Ρολάν, εσείς τώρα. Σύντομα, ναι. Το πρώτο ατού που έχουμε και το εξήγησε προηγουμένως ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είναι η συμμετοχή των ΜΕΝ και των ΔΕ στα διακυβεύματα για να γίνει κάτι το οποίο είναι ουσιώδες για την υγεία των εργαζομένων και βεβαίως και για την υγεία των επιχειρήσεων. Από την άλλη μεριά, δεύτερο στοιχείο, πράγματι επιθυμούμε να γίνει η εναρμόνιση αυτή για να αποφευχθούν στρεβλώσει του ανταγωνισμού στην βάση τη προστασία τη Υγεία. Θα είναι το χειρότερο πράγμα αυτό που μπορούσε να συμβεί. Να ληφθούν βεβαίω υπόψη οι πραγματικότητε των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Με την έννοια όμω ότι οι εργαζόμενοι του χρειάζονται την ίδια προστασία με αυτού των μεγάλων, αλλά βεβαίω να ληφθούν υπόψη και οι ικανότητε προσαρμογή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στις ε, νέες συνθήκες για το καύσιμο diesel. Τώρα είναι σαφές ότι δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η συζήτηση αυτή εδώ. Η μια συζήτηση όμως πρέπει να γίνει. Δεν ξεκινούμε από το μηδέν. Προχωρεί η νομοθεσία, για παράδειγμα στη Γερμανία αλλά και στην Αυστρία ή στις κάτω χώρες. Και ο σχετικός προβληματισμός είναι γνωστός. Όλοι αναγνωρίζουν ωστόσο ότι υπάρχει πρόβλημα τοξικότητας των ε, αναθυμιάσεων diesel ή των εξατμίσεων ε, diesel. Και χρειάζεται να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ένα τελευταίο. Μιλήσατε πριν για τη συμφωνία Νέψη και η κυρία Μακεντάιρ το Η σημασία της πρωτοβουλίας που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις και οι τομείς. Νομίζω ότι η συμφωνία Νέψη είναι ένα καλό παράδειγμα εν προκειμένου που μπορεί να ενταχθεί και μέσα σε αυτήν την κατηγορία της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων καθώς και της επιθυμίας να προχωρήσουν οι κοινωνικοί εταίροι και μάλιστα να προηγηθούν της νομοθεσίας. Και συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία ευθύνης των κοινωνικών επιχειρήσεων, των, μάλλον κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την νομοθεσία. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία μπορούν να επιτρέψουν ενδεχομένω να προχωρήσει η νομοθεσία, να βελτιωθεί, mm. αλλά δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας. Πάντως, ανυπομονώ, όχι απλά να αρχίσω διότι συνεχίζουμε άλλωστε την εργασία που έχουμε αρχίσει με την πρώτη δέσμη, αλλά θα συνεχίσουμε μετά από τον πρώτο γύρο. Θα έχουμε λοιπόν και περαιτέρω εμπειρίες στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε και νομίζω η προσπάθειά μας θα αυξηθεί σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά της. Ευχαριστώ κύριε Ρολάν, ευχαριστώ και τα υπόλοιπα μέλη που συμμετέσχουν στην συζήτηση και όπως έγινε σαφές νομίζω ότι σημαντικό είναι και το χρονοδιάγραμμα γιατί πρόκειται για την διάσωση ζώων αλλά βεβαίως και για την υλοποίηση από πλευράς επίπεδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι έχουμε τη δυνατότητα να λάβουμε αποφάσεις για τις προτάσεις αυτές και όπως είπε βεβαίως προηγουμένως και ο κύριος Όλσον αυτές οι προτάσεις θα γίνουν αρχές του 2019 και αν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε αυτά αρχές του 2019 τότε μπορούμε να στραφούμε και καλύτερα στους Ευρωπαίους πολίτες και ψηφοφόρους να εξηγήσουμε ότι πρόκειται για μια, ειδού κάνουμε μια προσπάθεια να υλοποιήσουμε αποφάσεις που θα βελτιώσουν τη ζωή των απλών ανθρώπων. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και μια πολυθετική ε, δήλωση μετά από αυτή την εντατική συζήτηση. Επομένως, 21-22 Φεβρουαρίου την επόμενη φορά που θα συζητηθεί αυτό στην Επιτροπή Απασχολήσεως. Τώρα, το υπαριθμό 6 της ημερήσιας διάταξης. Σύσταση του Συμβουλίου για τις ε, περιόδους άσκησης. Προβλέπω μάλιστα να ομιλήσω εγώ, από ό,τι βλέπω από τις σημειώσεις εδώ. Αλλά μια στιγμή να δω αν θα πρέπει να αρχίσω. Ως εξής. Στις 5 Δεκατού δημοσιεύθηκε η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση του Συμβουλίου για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ε, πρακτικές ασκήσεις ποιότητας. Ως συνέχεια της New Skills Agenda for Europe το 2016. Ο στόχος εν προκειμένου είναι να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τις ασκήσεις αυτές, για τις περιόδους δηλαδή ασκήσεως, σε μια κοινή συμφωνία σε ό,τι αφορά την ε, αποτελεσματικότητα και ποιότητα των πρακτικών αυτών εκπαιδεύσεων κάθε τους ασκήσεων και η σύσταση περιλαμβάνει και τα κριτήρια μαθήσεως καθώς και εργασίας των προσώπων αυτών με έγγραφες συμβάσεις το τι, ποια παιδαγωγική ε, στήριξη θα δοθεί αμοιβή ή αποζημίωση ή και αποζημίωση καλύτερα κοινωνική προστασία και άλλες ε, συνθήκες για την εκτέλεση αυτών των πρακτικών ασκήσεων. Η δε σύσταση περιλαμβάνει και ορισμένα κριτήρια για τις συνθήκες πλαίσια, όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο, την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, επιχειρήσεων, ε, εύκαμπτες προσεγγίσεις και κριτήρια ποιότητας. Έχουμε ορισμένους εδώ που ενδιαφέρονται για την σύσταση αυτού του Συμβουλίου. Σε ποιον μπορώ να δώσω το λόγο, στον κύριο Σόγκορ. Ορίστε, έχετε το λόγο κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Ένα καλό σύστημα και καλά σχεδιασμένο σύστημα δηλαδή για πρακτικές για πρακτική άσκηση νέων επαγγελματιών είναι σημαντικό γιατί μπορεί να τους επιτρέψει να περάσουν την επαγγελματική ζωή και πάντως προσφέρουν αξία και στους εργοδότες διότι έτσι μπορούν να εξεύρουν ε, προσοντούχα άτομα. Από κάθε άποψη λοιπόν οι ασκήσεις αυτές βελτιώνουν την παραγωγικότητα και την απασχολησιμότητα. Είναι σημαντικό να τονιστεί επίσης ότι χώρες που έχουν παράδοση σε, αυτές τις, ε, σε αυτή την πρακτική άσκηση αποδείχνουν ότι είναι και οι πιο ανθεκτικές στην οικονομική κρίση. Χρειάζεται να προωθηθούν λοιπόν τέτοια συστήματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θεωρούμε ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο την σύσταση αυτή του Συμβουλίου. Εδώ έχουμε ξεκινήσει καλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο. Η Γραμματεία έχει κάνει μια επισκόπηση των πιο σημαντικών θεμάτων που θα πρέπει να μας απασχολήσουν για να υπάρξει μια κοινή κατανόηση για το τι σημαίνει πρακτική άσκηση ποιότητας. Από δε το σχέδιο ψηφίσματος θα τονίσω ιδίω την ανάγκη διευκόλυνση συνεργασίας μεταξύ των αρχών των κροτών μελών, κοινωνικών εταίρων και άλλων προσφέρουν ε, πρακτική άσκηση, να υπάρχει ένα σύστημα παρακολούθησης για την ε, ε, ποιότητα διότι ενδεχόμενε καταχρήσεις θα έχουν πολύ δυσμενή επίπτωση, να αρθούν οι μη αναγκαίοι περιορισμοί, να προστατευτούν και άνθρωποι οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται και να εμπλακούν καλύτερα και συχνότερα και οι εργοδότες. Υπάρχουν και ορισμένα θέματα όπου νομίζω ότι χρειάζεται μια περαιτέρω μελέτη και εγώ θα υποβάλω εκεί κάποιες τροπολογίες. Πρώτα, Υπάρχουν μεν προγράμματα πρακτικής εξάσκησης σε ορισμένες χώρες μέλη, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Αυτό φαίνεται από τα νούμερα. Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για το θέμα αυτό, η συμμετοχή σε τέτοιες πρακτικές αξίσεις ξεκινά από 5% στην Βουλγαρία και φτάνει τα 53% στην Αυστρία. Με 15% η δική μου χώρα βρίσκεται και αυτή σχετικά κάτω σε ό,τι αφορά την χρήση αυτής της δυνατότητας πρακτικών ασκήσεων θα πρέπει για αυτήν να λάβουν έξτρα χρηματοδότηση οι χώρες που υστερούν. Δεύτερο, οι εργοδότες παίζουν σημαντικό ρόλο για την πρόθεση τέτοιων προγραμμάτων, διότι ταυτόχρονα πρέπει να γίνει προσπάθεια να στηριχθούν οι εργοδότες για να συμμετάσχουν. Διότι έρευνες δείχνουν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σπανίως έχουν ενδιαφέρον να προσφέρουν πρακτική άσκηση σε ενδιαφερόμενα άτομα. Γι' αυτό πρέπει ε, να ενταθεί η ενημέρωση για τα ωφέλη που προσφέρουν οι πρακτικές αυτές ασκήσεις, να δοθεί η χρηματοδοτική στήριξη και να μειωθεί η υπερητή γραφειοκρατία. Τρίτο, δεν υπάρχουν συγκρίσιμα δεδομένα για την ε, εφαρμογή των πρακτικών ασκήσεων αν υπάρξουν, θα υπάρξει και καλύτερη δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων. Και γι' αυτό αυτό οφείλει να γίνει. Τέταρτο, άλλο σημαντικό θέμα θα είναι να ενθαρρυνθούν προγράμματα πρακτικών ασκήσεων που να αφορούν και ανθρώπους οι οποίοι υστερούν είτε κοινωνικά είτε έχουν δυσκολίες μαθήσεως. Υπάρχουν τέτοια καλά παραδείγματα σε Γερμανία και Αυστρία για ανθρώπους με ιδιαίτερες ανάγκες. Τέτοια παραδείγματα λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες χώρες μέλη. Τα λέω όλα αυτά. Αναμένω βεβαίως να ε, συνεργαστώ και με τους υπολείπους ενδιαφερομένους για το θέμα αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Σόγκορ. Και τώρα από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, ο κύριος Λόπες. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι η ε, δεν μπορούσε να είναι εδώ και Γκουτιέρης, αλλά μάλλον ο κύριος Γκουτιέρης δεν είναι εδώ, αλλά έχω συζητήσει μαζί του τα στοιχεία, την αξιολόγηση Άλλωστε έχουμε από κοινού αναλάβει την προετοιμασία αυτής τη υποφορική ερώτηση. Καταρχάς θέλω να πω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτή τη σύσταση θέλει να βάλει τάξη, να συμπληρώσει, να βοηθήσει έναν από τους ευάλωτου ε, τομεί τη αγορά εργασία. αυτού που είναι μεταξύ ε, των σπουδών και της ε, Αγορά εργασία, δηλαδή στου ασκούμενου αυτού που συμμετέχουν σε προγράμματα μαθητείας. Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτές οι πρακτικέ για τη μετάβαση στην αγορά εργασία βοηθούν ε, να έχει κανεί ουσιαστική, να αποκτήσει ουσιαστικέ γνώσει ε, και να του προσφέρει δεξιότητες, γνώσει, για να μπορέσει να προσφέρει κάτι παραπάνω και στην επιχείρηση που το έχει προσφέρει αυτή τη θέση, αλλά και να είναι αποτελεσματική αυτή η μαθητή για να μπορεί να ενταχθεί μετά στην αγορά εργασία. Η δική μα πολιτική ομάδα δεν βλέπει τίποτε αρνητικό στη σύσταση, σε ό,τι το περιεχόμενο. Από γενική πλευρά όμω, αυτό που βλέπουμε να λείπει είναι συγκεκριμένα να αναφέρεται πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι της σύστασης. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για το ποιο είναι το εργαλείο ε, που θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν για την ε, συμμετοχή σε αυτό το τομέα. 153-167 είναι τα άρθρα ε, που, στα, οποία βασίζονται, στα οποία βασίζεται αυτή η σύσταση. Επίσης, μπορεί να προταθούν και άλλα εργαλεία, άλλου είδου εργαλεία από την Κομισιόν. Ξέρουμε ότι τα τελευταία 3,5 χρόνια συστάσεις υπήρξαν και αρκετές και όχι μόνο για αυτό το θέμα αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς πάντα για ευάλωτους ε, συνανθρώπους μας όπως είναι μακροχρόνια άνεργοι Παραδείγματο χάρη, έχουμε μα είχε απασχολήσει στην Επιτροπή μα το θέμα πολλέ φορέ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι έχει λάβει και κάποιες ε, αποφάσεις ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εργαζόμενοι αλλά και μαθητές είναι τα άτομα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούν να έχουν αυτό το διπλό στάτους, το διπλό καθεστώς αυτοί οι άνθρωποι για να μπορούν να έχουν και μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνάπτουν τις επιχειρήσεις. Επίσης, η αρχή της επικουρικότητας που πάντοτε περιλαμβάνεται σε αυτό το είδος τα κείμενα και είναι και μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία ή ως πρόσχημα για τη μη ρύθμιση τομέων που το επιτρέπουν οι συνθήκες. Για να υπάρχει μια νομική ισχύ. Εμείς θέλουμε να υπάρξει συμπληρωματικότητα και στο νομοθετικό κομμάτι. Τρίτον, θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Έχουμε τη σύσταση του 2014 για ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις ε, πρακτικές ε, για τις περίοδους ε, πρακτικής άσκησης. Τι μάθαμε, τι μάθαμε από αυτές τις ε, εμπειρίες, τι λειτουργήσε, τι δεν λειτουργήσε, γιατί μοιάζουν αυτά τα δύο. Γιατί αν συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε το ίδιο εργαλείο για τη ρύθμιση ενός ευάλωτου τομέα όπως αυτός, θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα αν λειτουργεί ή όχι αυτό το εργαλείο τελικά. Και τέλος, η πρόταση σύσταση συσχετίζεται και με την εφαρμογή του κοινωνικού πυλώνα. Ξέρετε βέβαια ότι η δική μας ομάδα είναι προσιλωμένη σταθερά ε, στον κοινωνικό πυλώνα. Προκύπτει όμως και εδώ το ίδιο θέμα. Ο κοινωνικός πυλώνας για μας πρέπει να είναι ένα εργαλείο, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και τα χρηματοοικονομικά, ε, ρυθμιστικά στοιχεία και εργαλεία στη συνέχεια. Και υπάρχει φόβος και κίνδυνος μήπως τελικά έχουμε μια απλή λίστα, έναν απλό κατάλογο συστάσεων για τις δημοσίες υπηρεσίες ή για την επαγγελματική παιδεία στην κατάρτιση, αλλά τίποτα παραπάνω. Ευχαριστούμε και τώρα λόγο στην κυρία Τρεμπέζιους από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή βεβαίως με τον οποίο θα συμφωνήσω τουλάχιστον εν μέρη, διότι πράγματι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανεργία των νέων είναι σε χαμηλά επίπεδα στις χώρες εκείνες που έχουν αυτό το διπλό εκπαιδευτικό σύστημα και μιλήσατε πριν για Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία και Δανία. Δεν ξέρω αν είναι σκόπιμο πράγματι να εξαχθούν τέτοιου είδους μοντέλα για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα στις χώρες που πλήγονται ακόμα σήμερα από την κρίση, παρόλο που εμείς θεωρούμε ότι είναι μια λογική προσέγγιση και θα θέλαμε να την υποστηρίξουμε. Όμως δεν είναι και για μένα απόλυτα βέβαιο πώς μπορεί να επιτύχει τον στόχο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι δεν είναι και αρκετά σαφής και η σύσταση του Συμβουλίου. Για μένα το πρόβλημα δεν είναι οικονομικό. Λέει για παράδειγμα μέσα καλά δομημένα προγράμματα πρακτικής εξάσκησης ε, ωφελούν και τους εργοδότες και τους εργαζομένους. Ταυτόχρονα μιλεί και για ποιότητα της άσκησης αυτής. Ναι, σωστά είναι αυτά τα πράγματα, αλλά είναι και λίγο ευχολόγια. Ίσως αυτό να γίνεται σε κάποια πιο απλά επαγγέλματα, όπως ας πούμε στο εξωτερικό εμπόριο ή στην προσφορά υπηρεσιών. Αλλά σε άλλα απαιτητικά επαγγέλματα, σε προσόντα κλπ. Δεν είναι και τόσο απλό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από τη δική μου χώρα παροιμήν η τεχνική εκπαίδευση είναι σε τρεις βαθμίδες. Αφενός δηλαδή η επιχείρηση παίρνει κάποιον, τον εκπαιδεύει, του δίνει ένα χαρτί στο τέλος, ένα δίπλωμα δηλαδή, κάτι το οποίο βεβαίως σημαίνει για την επιχείρηση απλώς μια επένδυση. Μπαίνει μετά στη δεύτερη βαθμίδα, είναι δηλαδή ε, πλέον εκπαιδευόμενος, ο οποίος ακόμα δεν μπορεί ωστόσο, σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, ε, να δημιουργήσει δική του αυτοτελή επιχείρηση. Και μετά έρχεται η τρίτη βαθμίδα, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος προχωρεί, περνάει την τελική εξέταση, γίνεται πλέον ε, τεχνίτης με πλήρη δικαιώματα αυτό βεβαίω όμω είναι πολύ ελκυστικό πλέον, να προσλάβουν τέτοια πρόσωπα δηλαδή, και οι επιχειρήσεις, διότι με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποσβέσουν την επένδυση που έχουν κάνει στην εκπαίδευση του παιδιού αυτό από την αρχή. Εάν όμως τώρα τη δεύτερη βαθμίδα μπορεί ε, ο εκπαιδευόμενο δηλαδή να δημιουργήσει δική του επιχείρηση, τότε δεν είναι πλέον συμφέρον για την επιχείρηση να του πληρώσει την αρχική του εκπαίδευση, διότι αυτομάτως αποκτά έναν ανταγωνιστή. Πρόκειται για έναν επιχειρηματικό κίνδυνο δηλαδή, τον οποίο θέλω να επισημάνω εδώ στον εισηγητή. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να ψάξουμε να βρούμε κάποιες ευφυείς λύσεις, ώστε να μπορούν ας πούμε, οι επιχειρήσεις να συμμετέχουν οικειοθελώς ή εν πάση περιπτώσει οι χώρες μέλη στην βάση της οδηγίας να έχουν ε, επαρκή ευχέρεια επιλογής ώστε να μην υπάρξει ανατροπή στις ε, αγορές εργασίας τους και μετά όπως είπε και ο κύριος Λόπες ότι η αγορά εργασίας είναι βεβαίως εθνική αρμοδιότητα και πρέπει να παραμείνει και γι' αυτό και η πολιτική μας ομάδα δεν δέχεται παραβίαση της αρχής αυτής γι' αυτό θεωρούμε ότι η οδηγία πρέπει να παραμείνει μη δεσμευτική με αυτή την έννοια η πολιτική μου ομάδα των ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών υποστηρίζει την ε, πρόταση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο σε εκπρόσωπο της ομάδας Άλντε, των φιλελευθέρων. Αν δεν βλέπω κανένα να είναι παρόν. Η κυρία Χάρκιν δεν είναι παρούσα. Κανείς νομίζω δεν την αντικαθιστά. Καλώς. Τώρα, από την ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς, η κυρία Γκονζάλες Πένιας. Ναι, ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Θέλω να ευχαριστήσω ε, την εισηγητρία για την προφορική ερώτηση και το ψήφισμα, την πρόταση ψηφίσματο. Έχουμε πολλά κοινά σημεία. Συμφωνούμε ε, εν γέννη με τι ερωτήσει προς το Συμβούλιο και με την γενική αντίληψη σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, το έχουμε ξαναπεί. Θεωρούμε ότι οι νέοι που υποφέρουν εδώ και μια δεκαετία από την υποβάθμιση των συνδικών εργασίας πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο προστασίας ώστε να προλάβουμε να αποτρέψουμε αυτά τα συμβόλαια, αυτές οι συμβάσεις να γίνουν επισφαλείς θέσεις εργασίας. Έχουμε και τροπολογίες ε, να καταθέσουμε σε τέσσερα σημεία Πρώτα απ' όλα την μετάβαση από τον χώρο της εκπαίδευσης ε, στην αγορά εργασίας. Αυτά τα συστήματα μαθητείας θα πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό στόχο τη μετάβαση από τις σπουδέ ε, στην αγορά εργασίας και πρέπει να υπάρχει σταθερότητα στην θέση εργασία που θα δεθούν. Σε κάποιες χώρες Υπήρχε αυτή η σύμβαση μαθητείας ε, ορισμένου ε, χρόνου, όμως λόγω των διαδοχικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που απορρίθμισαν ε, την αγορά εργασίας σε πολλές χώρες έχει ανοίξει αυτή η πόρτα που επιτρέπει το να διονίζονται αυτές οι συμβάσεις μαθητείας. Οπότε έχουμε κακοπληρωμένους εργαζόμενους τελικά και όχι μαθητευόμενους. Επίσης ό,τι αφορά τα ποιοτικά προγράμματα μαθητείας. Ο σε μια προηγούμενη έκθεση του λέει ότι θα πρέπει να έχουμε κανόνες ποιοτικού ε, για τους μαθητευόμενους ε, για να μην καταλήξουν αυτοί να εργάζονται εργάζονται σε χαμηλής εξειδίκευσης θέσεις εργασίας. Θέλουμε να υπάρχει ένας χάρτης για να βλέπουμε ε, πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι πρακτικές. Ε, υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία, η Γερμανία που είναι επιτυχής όλη αυτή η διαδικασία, αλλά σε άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, ε, εκεί βλέπουμε συχνά αυτά τα μέτρα να μην οδηγούν ε, στην κατάληψη μιας θέση εργασία, αλλά διατηρούν ε, σε μόνιμη επισφάλεια και αβεβαιότητα τους νέου, Δηλαδή αντικαθιστούν θέσεις σταθερέ με αυτές τι επισφαλεί θέσει εργασία. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα ποιοτικό πλαίσιο για αυτές τις περιόδους ε, άσκησης ή μαθητείας. Να υπάρχει γραπτή σύμβαση, να καθορίζεται δε και η αμοιβή, οι απολαβές. Σε ό,τι δε αφορά την αποζημίωση, θεωρούμε ότι θα μπορούσε να είναι επιτυχής αυτή η διαδικασία, αλλά θα πρέπει να συμμετέχει αγορά εργασίας. Χρειάζεται λοιπόν χρηματοδότηση ε, και θα πρέπει να υπάρχει και επαγρύπνηση για να μην υπάρχουν ε, περιπτώσεις εκμετάλλευσης των νέων. Τέλος, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και τους τελικούς στόχους, θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τι απαιτούμενε αναφορές στην Ήπεθρο, στις αγροτικές περιοχές. Θα πρέπει επίσης να αναφερθούν τα άτομα με αναπηρία και να τεθούν οι βάσεις ώστε να λαμβάνει υπόψη η ισότητα των δύο φύλων. Οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να παρακολουθείται ο οργανισμός αυτός, ε, να να, ώστε να ελέγχονται αυτά τα προγράμματα. Και με το ψήφισμά μας θα πρέπει να φροντίσουμε να έχει θετικές επιπτώσεις αυτό το πρόγραμμα και να μην οδηγεί σε εκμετάλλευση και επισφάλεια. Ε, thank Σας ευχαριστώ από τους Πρασίνους, η κυρία Ράιντκε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα πήγατε πάρα πολύ γρήγορα αυτή τη φορά όλα τα θέματα και δεν πρόλαβα την αρχή τη συζήτηση. Τέλο πάντων, μιλάμε για το πλαίσιο για αποτελεσματικέ και ποιοτικέ περιόδου άσκηση. Εδώ νομίζω ότι πρέπει να εισάγουμε κάτι που να λειτουργεί ω πλαίσιο αναφορά μεταξύ των κρατών μελών για τι περιόδου ε, μαθητεία και τα πρότυπα για αυτά. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί τα τελευταία χρόνια είδαμε τέτοια μεγάλη ποικιλομορφία των ασκήσεων και μαθητών μεταξύ των μελών, που δεν είναι απλώ δύσκολο οι σταζιέροι να πάνε από το ένα κάτω μέλο στο άλλο, αν θέλουν διασυνοριακή εμπειρία, αλλά επίση κάποιε φορέ γίνεται πολύ δύσκολο να ε, υπάρξουν συγκρίσιμα δεδομένα οι διαφορετικέ πρακτικέ, δηλαδή να συγκριθούν μεταξύ του. Μάλιστα, σε κάποια κάτι μέλη υπάρχει εκμετάλλευση ιδίω των νέων ονομάζονται ασκήσεις ή μαθητείες, πράγματα που δεν είναι κάτι τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ποιότητα. είναι σημαντικό αυτό. Και θα πρέπει τα πρότυπα να ακολουθούν από όλα τα κάτι μέλη όταν μιλάμε για περίοδους άσκησης. Λόγω χάρη η αμοιβή θα πρέπει να είναι ένα στοιχείο. Θα πρέπει να πληρώνονται οι ασκούμενοι, να υπάρχει ένα ε, συμβόλαιο με νομική ισχύ. Οι ασκούμενοι να μην είναι εκεί ως ε, χαμηλόμιστοι ε, στο εργατικό δυναμικό, αλλά κάτι να μαθαίνουν για τη δουλειά τους στην ουσία. Είναι λοιπόν μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το διάστημα, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ακαδημαϊκή εκπαίδευση και η περίοδοι άσκηση βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Κάποια κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση ω πιο αξιόλογη και πολύτιμη για την κοινωνία ε, εξορισμού. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε περισσότερο βάρο στι ε, περιόδου άσκηση για να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Και επίση ένα σημείο που ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, θέλω να το επαναλάβω και εγώ, πρέπει ο κόσμο των επιχειρήσεων και εταιρείων να παίξει ένα ρόλο. Το θέμα του κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση ω αγορά θα είναι επιτυχή και στο μέλλον θα εξαρτηθεί από το πόσο ε, υψηλά προσόντα και ε, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον θα έχουν οι μελλοντικοί μα εργαζόμενοι οι επιχειρήσεις ακόμη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για, την, για το να επενδύσουν, στο να βεβαιωθούν ότι υπάρχει τέτοιο εργατικό δυναμικό, ποιοτικό και ικανό και στο μέλλον. Το να επενδύσουμε στην ποιότητα και τι αποτελεσματικέ λοιπόν περιόδου άσκηση θα είναι ένα πολύ σημαντικό σκέλο όλη αυτή τη προσπάθεια. Εκεί πρέπει να αναλυθεί ευθύνη από τι επιχειρήσει και τι εταιρείε. Γι' αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να δηλωθεί ότι κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτόν τον τομέα. Ακόμη και αν κάτι του κοστίσει χρηματικά, τα χρήματα αυτά τουλάχιστον θα είναι επενδύσει που θα τι αποσβέσουν στο μέλλον. Ευχαριστούμε. Και τώρα από την EFTD δεν έχω κάποιον στον κατάλογό μου. Κανείς από την ΕΝΕΦ. E Ίσως κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Παρακαλώ. Λάβετε το λόγο, κυρία Μπάχου. Ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζουμε την ε, μελέτη της πρωτοβουλίας αυτής από το Ευρωκοινοβούλιο εγώ ίσως απλώς να τονίσω ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει πολύ θετική ε, απόκριση ως τώρα από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων. Από την ημερομηνία της θέσης σε ισχύ της πρότασης θα γνωρίζετε ότι όλοι οι κοινωνικοί εταίροι, εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν καλωσορίσει αυτή την πρωτοβουλία. Βεβαίως υπήρξαν και κάποιες προτάσεις για προσθήκη σε σχέση με την πρόταση στο περιεχόμενό της, αλλά αυτό είναι κάτι αναμενόμενο. Το περίμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως θα ξεκινήσουν τώρα και διαπραγματεύσει εντός του Συμβουλίου. Να πω ότι βασίζεται η πρωτοβουλία αυτή στην πολλή δουλειά που έγινε, στην, ε, στο συνασπισμό για τις περίοδους άσκησης, μια πρωτοβουλία όπου υπήρχαν ένα σωρό ενδιαφερόμενοι, κοινωνικοί εταίροι, κράτη-μέλη, επιμελητήρια, ενώσεις και σύλλογοι και Ακόμη πιο πρόσφατα ήδη οι ασκούμενοι, οι ίδιοι σταζιέρ. Διότι πέρσι προβλέπα, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο ασκουμένων τη Ευρώπη, ώστε να μπορούν και αυτοί να κάνουν τη φωνή του να ακουστεί στο επίπεδο τη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικών. Να δώσουν προσανατολισμού και κατευθύνσει για να προστατευτούν τα δικαιώματά του. Ω προ το περιεχόμενο τη πρόταση, ίσω λίγα λόγια, εάν μου επιτρέπετε, προσπαθήσαμε να καλύψουμε δύο διαφορετικά επίπεδα παρέμβασης καθορίσαμε τέσσερα σύνολα κριτηρίων που επικεντρώνονται στο ίδιο το σύστημα των ασκήσεων και μαθητιών από την πλευρά του εκπαιδευομένου, του ασκούμενου. Ποια, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να ισχύουν για να είναι επιτυχής η περίοδος της άσκησης, να είναι μια επιτυχημένη παιδαγωγική εμπειρία. Είδαμε λοιπόν το σκέλος το μαθησιακό αλλά και την ε, διάδραση που χρειάζεται να υπάρχει εδώ. Συνεργασία δηλαδή μεταξύ των εταιριών ως χώρο μάθησης και της επαγγελματικής κατάρτισης ε, στα σχολεία, τις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης. Υπάρχει αμοιβαία ανάγκη παρακολούθησης και στα δύο επίπεδα, τα δύο σκέλη, για να βεβαιωθούμε ότι η περίοδος άσκησης και ο ασκούμενος στο τέλος παίρνει ένα συνδυασμένο σύνολο παιδαγωγικών ε, διδαγμάτων που να το χρησιμεύουν και για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων του και για την επαγγελματική του σταδιοδρομία στο μέλλον. Υπάρχει επίσης το θέμα της αμοιβή ε, αποζημίωσης έστω με κοινωνικό χαρακτήρα καθώς και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Είναι και αυτά στοιχεία που θα πρέπει να ισχύουν, να παρέχονται βάσει των εθνικών προτύπων και της εθνικής νομοθεσίας. Το δεύτερο σύνολο κριτηρίων αφορούν τις προϋποθέσεις πλαίσια, διότι οι περίοδοι άσκησης δεν ισχύουν, εν κενό είναι μέρος του γενικότερου συστήματος επαγγελματικής ε, κατάρτισης και εκπαίδευσης. Οπότε θεωρούμε ότι για να είναι επιτυχής η περίοδοι άσκησης και μαθητείας και να είναι και ποιοτικέ, θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο το τοπίο, ένα συγκεκριμένο σύστημα, ένα ρυθμιστικό δηλαδή πλαίσιο που ευθύ εξ αρχή να ορίζει τι υποχρεώσει των ε, διαφόρων εμπλεκομένων σε αυτή τη διαδικασία. Εδώ υπάρχει σημαντική συμμετοχή και των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και την παροχή και την υλοποίηση των, ασκήσεων των περίοδων άσκηση, αλλά κάτι που το έθιξαν και οι βουλευτές της παρεμβάσης τους, πολύ σημαντικό, είναι η αναγνώριση η αναγνώριση των περίοδων άσκησης ως ενός πολύτιμου, ε, μιας πολύτιμης διαδρομής ε, για την απόκτηση εμπειρίας. Είναι σημαντικό για το σύστημα των επαγγελματικών προσώπων και να αναζητήσει κανείς ε, οριζοντίως ή σε υψηλότερο επίπεδο και άλλες επαγγελματικές ευκαιρίες ή αποκόμιση επαγγελματικών προσόντων. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της πρότασης είναι οι συστημικές προϋποθέσεις. Κοινώς η στήριξη. Οικονομική ή μη οικονομική στήριξη στις εταιρείες μικρομεσαίες ιδίω για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας περιόδους άσκησης και να γίνουν ένα μαθησιακός χώρος με ποιότητα. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βρείτε και συστάσεις προς τα κρατημέλη ως προς το τι εξακολούθηση θα πρέπει να δοθεί στην υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε ότι ενδεχομένως ως προς το κείμενο της σύστασης να είναι εύκολα επιτευχθεί πολιτική συμφωνία. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτή η πολιτική συμφωνία να λάβει σάρκα και οστά σε εθνικό επίπεδο. Να υλοποιηθεί και σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις που γύρει πρόταση από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα είναι να τη στηρίξη να προσφέρουμε στην υλοποίηση καθώ και την δημιουργία υπηρεσιών για την υποστήριξη των, ασκήσεων, των περιόδων άσκηση. Αυτό θα το, το είδαμε και την εβδομάδα σε σχέση με τα στάζια και τι περιόδου άσκηση που έγινε στη Βιέννη τον Νοέμβριο. Εβδομάδα για το θέμα αυτό συγκεκριμένα. Από δική μου πλευρά, αυτά προ στιγμή. Είμαι στη διάθεσή σα για απαντήσει. Ευχαριστούμε που ήρθατε και μας δώσατε αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πληροφορίες, χρονοδιάγραμμα της πρότασης. 5η ναι, αυτή τη Πέμπτη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 25 Ιανουαρίου στι 12 το μεσημέρι. και η έγκριση στην Επιτροπή Απασχόλησης της 27 Φεβρουαρίου. Η έγκριση στην Ολομέλεια, στην Ολομέλεια του Μαρτίου. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ερμηνεία και εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Έχουμε ένα πρόβλημα. Διότι η κυρία Μακιντάιρ, που είναι η συντάκτρια της γνωμοδότησης αυτής, έχει πάει σε μια άλλη επιτροπή. Άρα απουσιάζει αυτή τη στιγμή. Και δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να περάσουμε απλά στο επόμενο θέμα, γιατί το επόμενο θέμα είναι ακρόαση υποψηφίων. Και δεν ξέρω καν αν έχουν έρθει. Οπότε, τι να κάνουμε, μήπως να δώσουμε το λόγο στους κλάδες συγκητές. Και όταν έρθει η κυρία Μακεντάρη να πάρει αυτό το λόγο, έρχεται τρέχοντας. Έρχεται σε 10 λεπτά μάλιστα. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Είμαστε... Έχουμε προχωρήσει αρκετά, αλλά αν κάνουμε διάλειμμα θα φύγουν οι ορισμένοι συνάδελφοι που είναι εδώ, ενδεχομένως. Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε περιμένοντας την κυρία Μάκιντάιρ και να δώσουμε το λόγο σε έναν δυο σκιώδους εισηγητές. uh, on, uh, this item. Για το θέμα αυτό λοιπόν θα ήθελα καταρχάς να δώσω το λόγο στην κυρία Σαντέρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω η συγγήτρια να ενημερωθεί κάποιος να τις μεταφέρει τις πληροφορίες και τα σχόλιά μας ε, για την ε, γνωμοδότηση που μας προτείνει σήμερα προς Θέλω να την ευχαριστήσω για αυτό το σχέδιο γνωμοδότης πρώτα απ' όλα. Ένα κείμενο που κατά την άποψή μου είναι μια πολύ καλή βάση εργασίας για την ομάδα μας. Θα καταθέσουμε βέβαια ορισμένες τροπολογίες για να συμπληρώσουμε το κείμενο σε κάποια σημεία που θα σας αναφέρω Αφού υπάρχουν δε αρκετοί απόντε, ελπίζω να έχω και πιο πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, εφόσον είμαστε και μπροστά στο χρονοδιάγραμμα. Σε ό,τι αφορά την πρώτη παράγραφο τη γνωμοδότηση τη κυρία Μάκεντάρη, νομίζω ότι σημαντικό θα ήταν το φάσμα να το ε, διευρύνουμε, σε ό,τι αφορά δηλαδή τα καινοτόμα στοιχεία που θεωρούμε ότι αποτελούν πρόοδο. Αναφέρει ορισμένα το σχέδιο γνωμοδότησης ε, εστιάζει στην απλούστευση κυρίως, στη ρυθμιστική απλούστευση και στην μείωση του διοικητικού φόρτου, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Φυσικά και αυτό είναι σημαντικό. Αποτελεί προτεραιότητα όμως η νομοθετική ε, δράση δεν περιορίζεται σε αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε και τη νομοθετική διαδικασία και να ζητήσουμε να υπάρχει διοργανική συνεργασία σε βάθος και ενίσχυση της διαφάνειας αυτής της νομοθετικής διαδικασίας. Πάντοτε σε σεβασμό προς την αναλογικότητα και την επικουρικότητα. Ένα αυτό. Δύο. Το 2 μιλά για τον προγραμματισμό των εργασιών. Η Διοργανική Συμφωνία προτείνει σημεία τα οποία συνιστούν πρόοδο στον τομέα αυτό και με τα οποία Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα αποκτήσουν έναν σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την εκπόνηση των προγραμμάτων εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κείμενο θα ζητήσει περισσότερη διαφάνεια, Το πάντων θα θεσπίσει περισσότερη διαφάνεια και θα υπάρχει αυτή η υποχρέωση νόμιμης και θεμητής συνεργασίας. Στην, στις επόμενες παραγράφους γίνεται λόγος για το Small Business Act, προτεραιότητες μικρές επιχειρήσεις, αυτή η αρχή. Νομίζω ότι πράγματι και Κοινοβούλιο και Συμβούλιο αλλά και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνουν περισσότερα ώστε να δίνεται προτεραιότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας. Νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν το 99% υπενθυμίζω του ε, επιχειρηματικού ιστού σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση αντικτύπου, το 5. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έπρεπε σε έναν κανονισμό να ορίζουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό μελών από το Κοινοβούλιο που θα είναι απαραίτητα για να γίνει μια αξιολόγηση αντικτύπου. Νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε πολύ περισσότερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τις δημόσιες διαβουλεύσεις και τις διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους. Euh, Νομίζω θα πρέπει να το συμπληρώσουμε λίγο παραπάνω αυτό το σημείο, τονίζοντας τη σημασία του και να πούμε ότι θα πρέπει τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων να τίθενται στη διάθεση των ε, μερών της διαβούλευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Παράγραφος 10. Εδώ γίνεται λόγος για τον καθορισμό στόχων για τη μείωση του φόρτου, του διοικητικού φόρτου. Εδώ θα ήθελα να αναφέρονται συγκεκριμένα πιο πολλά σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο και την ε, διαδικασία. Τέλος, ένα σημείο θέλω να αναφέρω, καταλήγοντας, είναι ένα σημείο που δεν περιλαμβάνεται στο σχέδιο γνωμοδότησης και το οποίο αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξης. Πιστεύω ότι πρέπει να μείνουμε στην σημασία ε, που έχει οι εμπειρογνώμονες Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να συμμετέχουν στην εκπόνηση των κατεξουσιοδότηση πράξεων, ώστε τα μηνύματα που θέλουν να περάσουν οι συνομοθέτες σε μια νομοθετική, βασική νομοθετική πράξη, να είναι πιο σαφή να μην παρερμηνεύονται. Και πρέπει να είναι πιο διαφανείς αυτές οι πράξεις. Καλό θα ήταν λοιπόν γι' αυτό να υπάρχει ένα κοινό μητρό για τις της πράξεις. Αυτά ήθελα να σας μεταφέρω, κυρία Πρόεδρε, ως μηνύματα προς την εισηγήτρια. Και θα είμαι ιδιαίτερως ευτυχής ε, να συνεργαστώ με όλους τους και όλους Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι βέβαια ότι κάποιος παίρνει σημειώσεις αναλυτικές για να ενημερώσει την κυρία Μακιντάιρ. Η κυρία Γιονγκέριους, Ζονγκέριους έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπρόντο Μπενιφάι ε, δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ που είναι ο σκιώδης ηγητής μας. Και δηλώνει ότι κολλείεται και έχει ένα σύντομο μήνυμα το οποίο σας διαβάζω. Και βεβαίως αποστέλει τους χαιρετισμούς του. Θέλει πρώτα να ευχαριστήσει τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης. Λέει ότι βεβαίως το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για την ορθή λειτουργία των θεσμών και του τρόπου εργασίας, αλλά και στην καθημερινό καθημερινή μας εργασία, δηλαδή απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις. Ως σκιώδης συγητής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών εκφράζει την ελπίδα ότι θα σημειωθεί σημαντική συνένεση, ο Μπραντ, να υπάρξει δηλαδή μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και να μπορέσουν να συμμετάσχουν όσοι ενδιαφέρονται για τους πολίτες της Ένωσης. Βεβαίως η βελτίωση της νομοθεσίας δεν σημαίνει απορρίθμιση. Θα πρέπει μάλλον να βασιστεί σε μια καλά συντονισμένη πολιτική που θα οδηγήσει σε βελτιωμένη ποιότητα η προστασία των εργαζομένων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης ή τον τόπο εργασία ή τον τύπο συμβάσεως. Θα πρέπει όλοι να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο οι εργαζόμενοι. Κατά την άποψή του το πρόβλημα συχνά εντοπίζεται στην ερμηνεία της νομοθεσίας που καμιά φορά είναι μονομερής. και δίνει και παραδείγματα. Δύο σημαντικούς φακέλους και για τη δική μας δουλειά δηλαδή που εξακολουθούν να τροχοπεδούνται στο Συμβούλιο. Αφενός για την ισότητα των φίλων στα διοικητικά συμβούλια που λέει τουλάχιστον 40% μη εκτελεστικών μελών του υπό αντιπροσωπευμένου φίλου στα διάφορα συμβούλια καθώς επίσης και τις ίσεις μεταχείρισης μεταξύ προσώπων, ανεξαρτήτως ε, φίλου, θρησκείας, ικανότητας ή ε, ε, αναπηρίας και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν σημαντικό να δώσουμε τη δυνατότητα στις προτάσεις αυτές να ξεφύγουν επιτέλους από το Συμβούλιο, από όσο προχωρήσουν δηλαδή και να γίνει μια προσπάθεια για διαφανή και αποτελεσματική νομοθεσία στον χώρο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Thank uh, Υπάρχει άλλος κανείς εκ των μελών που έχει συμμετάσχει, όχι. Α, η Γκαβριέλε Τσίμερ, πρόεδρος της Ενωτικής Αριστεράς. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Είχε από μακρού ανακοινωθεί ότι θα εγκύψουμε εμείς ως Επιτροπή Απασχόλησης στα θέματα των διεθνών συμβάσεων για την βελτίωση της νομοθεσίας και ούτω καθεξής. Έχουμε το σχέδιο τώρα γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής Απασχολήσεως και εξεπλάγει κάπως διότι στο όλο αυτό κείμενο δεν περιλαμβάνεται η συγκεκριμένη αξίωση για κοινωνική απασχόληση. Δηλαδή πρόκειται για μια γνωμοδότηση που θα μπορούσαν να είχαν συντάξει άλλε κοινοβουλευτικέ επιτροπές. Εμεί θα έπρεπε να αξιώσουμε συγκεκριμένα και ρητά να υπάρξουν κοινωνικές προδιαγραφές προστασίας. Και αυτό αρχίζω εδώ με την παράγραφο 10. Διότι, προφανώ ο εισηγητή θεωρεί ότι πρόκειται για κανόνες προστασίας των απασχολουμένων, που οι κανόνες όμω αυτοί αποτελούν βάρος, στα αγγλικά burden. Πώς να συμφωνήσω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να φροντίσουμε ειδικώ να μην σημαίνει η βελτίωση της νομοθεσίας ότι καταργείται η κοινωνική προστασία διότι δήθεν επιβαρύνει τις επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτό, πάνω σε αυτό θα πρέπει να το τοποθετηθούμε. Να πούμε δηλαδή πώς θα επιτύχουμε βελτιωμένη νομοθεσία υπέρ των εργαζομένων. Προστασία της εργασίας, δικαίωμα στην εργασία, δικαίωμα στην διαβούλευση. Η βελτιωμένη νομοθεσία δεν επιτρέπεται να οδηγήσει σε περιορισμό των δικαιωμάτων προστασίας των εργαζομένων. Αυτό είναι κρίσιμο για μένα για να μπορέσω να προσεγγίσω καν την πρόταση αυτή. Τονίζω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 μόνο στις μισές νομοθετικές προτάσεις είχε κάνει μελέτες αντικτύπου επικαλούμενη πάντοτε πίεση χρόνου. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Μεταξύ άλλων, επρόκειτο για έλλειψη μελετών αντικτύπου για κοινωνικά θέματα και για περιβαλλοντικά. Δηλαδή για τέτοιου είδους νομοθετικές προτάσεις. Αυτά όμως είναι κύρια σημεία που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έχουν ενταχθεί στην διαθεσμική συμφωνία. Τέλος, οι δημόσιες ακροάσεις είναι σημαντικές, δεν θα μπορέσουν όμως ποτέ να υποκαταστήσουν τον ε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο. Επιτρέψτε μου να αρκεστώ σε αυτά τα λόγια πρώτα. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να προχωρήσουμε στην κατάθεση τροπολογιών και να συζητήσουμε και μέσω αυτών πώς θα καταλήξουμε σε μια ενιαία θέση της Επιτροπής Απασχολήσεως. Ευχαριστώ. Thank you. And then we... Σας ευχαριστώ. Να που θα πάμε τώρα στο πρώτο όνομα του καταλόγου μας, την κυρία Μάκιντάιρ. Δεν είσαστε εδώ όταν ξεκίνησε η συζήτηση. Είμαι όμως βεβαία ότι τα επιχειρήματα τα γνωρίζετε λίγο πολύ. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο για να με συσάγετε το θέμα παρόλο που έχουν παρέμβει ήδη δύο ε, αγορητές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με συγχωρείτε που δεν ήμουν εδώ στην αρχή της συζήτηση. Ε, θα ήμουν εκεί και μισή. Ε, ήμουν στην ώρα μου δηλαδή, αλλά από ό,τι κατάλαβα ε, άργησα γιατί εσείς είχατε προλάβει νωρίτερα να ξεκινήσετε. Ήμουν σε δύο επίτροπε παράλληλα. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερο που έχουμε αυτή την ευκαιρία να συζητήσουμε τη Διοργανική Συμφωνία για την Καλύτερη Νομοθεσία και νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής αυτής το γνωρίζουν καλά. Είμαι ένθερμη υποστηρίκτρια της καλύτερης νομοθεσίας. Γι' αυτό πραγματικά θέλω να κάνουμε ό,τι μπορούμε από την Επιτροπή αυτή για να βεβαιωθούμε ότι η υλοποίηση της διοργανικής συμφωνίας δεν είναι μια ευκαιρία που θα πάει χαμένη. Υπάρχει μια σειρά από συστάσεις για το πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε λοιπόν τη συμφωνία και θεωρώ ότι είναι σημαντικό να έχουμε καλή νομοθεσία που να ορίζει το τι θα κάνουμε, είτε την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, την υγεία του, τη δημιουργία νόμων για καλύτερε θέσει εργασία. Νομίζω σημαντικό είναι η νομοθεσία να είναι όσο το δυνατόν πιο απλή και ε, εύκολο να ακολουθηθεί. Δεν πρέπει να κάνουμε συμβασμούς για τα πρότυπα στους νόμους που θεσπίζουμε, όμως πρέπει να είναι απλό ο κόσμος να καταλάβει και να μπορεί να τηρήσει τον νόμο. Πολύ συχνά βλέπουμε νόμο με ε, απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτό που θα ελπίζαμε να γίνει δηλαδή μέχρι τη στιγμή της ερμηνείας και της ε, θέσης εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο, δηλαδή προβλήματα και μπορώ να σας δώσω και παραδείγματα ε, αλλά δεν θα το κάνω για να μην χάσουμε και άλλο χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι η νέα διοργανική συμφωνία έχει πολύ ενδιαφέροντα και συναρπαστικά εργαλεία που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε. Πιο συγκεκριμένα ήθελα να αναφέρω την ετήσια έρευνα φόρτου. Πιστεύω ότι ένα από τα βασικά μηνύματα αυτής της Επιτροπής θα μπορούσε να είναι πώς θέλουμε η ετήσια έρευνα φόρτου να ε, εξελιχθεί και να εφαρμοστεί. Θα ήθελα να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται και η ετήσια έρευνα ανάπτυξη. Η Επιτροπή μα δηλαδή να απαντά ετησίω σε μια έρευνα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώ τα κράτη-μέλη μεταφέρουν, υλοποιούν και ε, τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Φυσικά, σε σχέση με τι αρμοδότητε τη Επιτροπή μα, εδώ θα είχε να κάνει με την νομοθεσία ε, για την εργασία και την απασχόληση. Μια τέτοια τήσια έκθεση θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για μα και του πολίτε μα, ώστε να δούμε την προστιθέμενη αξία τη ευρωπαϊκή νομοθεσία και να εκτιμήσουμε το κατά πόσον τα κράτη-μέλη την αξιοποιούν. Πολύ συχνά δηλαδή βλέπουμε την Ευρώπη να κατηγορείται για νομοθεσία που ήταν ουσιαστικά ε, μια χρυσή κορνίζα που εκμεταλλεύτηκαν τα κράτη-μέλη, χωρίς περιεχόμενο όμως. Λυπούμε που θα παραδεχτώ ότι αυτό ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω ότι μέρο των λόγων που πρότεινε το Ηνωμένο Βασίλειο και προτίμησε την αποχώρηση είναι γιατί λένε ότι υπήρχε σωρία νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια ε, και αυτό ενοχλούσε. Όμως πρόκειται απλώς για ένα ε, ιδανικό πλαίσιο που τελικά έφευγε από εδώ από εμά και κατέληγε να μην σημαίνει τίποτα όταν έφτανε στο κατόφλι μια μικρομεσαία επιχειρήση που η καημένη δεν μπορούσε να την ερμηνεύσει. Αυτό λοιπόν ω τα πρότυπα και τι μελέτε αντικτύπου οι μελέτε αντικτύπου δεν χρησιμοποιούνται παρκώς και θα πρέπει να είναι πιο προσβάσιμε. Πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που έχουν επιφυλάξει ω προ την ιδέα αυτή, αλλά υπάρχει ένα βασικό λόγο που θα ήταν πολύ υποφελής αυτέ οι μελέτε αντικτύπου, διότι ε, μπορούν να ενισχύσουν τη θέση μα στι διαπραγματεύσει των τριμερών διαλόγων. Το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή διεξάγει μία ε, ε, μελέτη αντικτύπου για την καλύτερη νομοθεσία, όμως καθυστερεί. Εάν είχαμε τη δική μα μελέτη που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και την προάσπιση των θεσεών μα. Δεν θα πρέπει να φοβούμαστε να κάνουμε μια μελέτη των επιπτώσεων των δικών μα τροπολογιών. Και θα μπορούσαν τέτοιε μελέτε να γίνουν και εξ ώστε τα προβλήματα να εντοπίζονται και να θεραπεύονται. Ένα άλλο ε, θέμα που ε, εντοπίζω είναι οι ενδιάμεσε διατάξει. Θυμίζουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αρμοδιότητά τη να απαντά στι εκθέσει μα ιδίας πρωτοβουλία. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει μία απάντηση και εξακολούθηση σε αυτέ τι ερωτήσει που να έχει νόημα. Καλωσορίζει επίση το γεγονό ότι η διοργανική συμφωνία αναγνωρίζει την ανάγκη οι μικρομεσαίε να υποστηριχθούν. Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι η ραχοκοκαλιά τη οικονομία μα και δημιουργούν το 90% των ένθεσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό η Επιτροπή μα να στηρίξει τα στοιχεία που περιλαμβάνει η διοργανική συμφωνία και θα βοηθήσουν τις μικρομεσαίες να τηρήσουν την νομοθεσία και ταυτόχρονα να κάνουν και την ε, ουσιαστική του δουλειά. Θα ήθελα λοιπόν, ενώ συνεχίζω την επισκόπηση όλων αυτών των στοιχείων, να πω ότι ανυπομονώ να ακούσω τις απόψει που δεν άκουσα ω τώρα. Ξέρω ότι υπάρχουν διαφορετικέ απόψει, αλλά η βοηθό μου κατέγραψε προσεκτικότατα τα σχόλια που έγιναν ω τώρα. Οπότε θα φροντίσω να ενημερωθώ και ανυπομονώ να ακούσω τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Εκ προσωπείτε εσείς τον Άλντε, δηλαδή την ομάδα των φιλελευθέρων, κύριε Καλβέτ. Ε, ναι, ευχαριστώ κυρία Ρόεδρε. Ο κ. Καβαντά είναι ο δικός μας και ο Με παρακάλεσε να αναγνώσω εξ ονόματός του σύντομο σχόλιο. Λέει λοιπόν ότι ευχαριστεί την εισηγήτρια για το σχέδιο Τη γνωμοδοτήσεω και κάνει και ορισμένα σχόλια. Πρώτο, χέρι για την διαθεσμική συμφωνία που διευκολύνει τι σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, η ετήσια έκθεση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την μείωση των βαρών καθώς και το ε, Συμβούλιο Παρακολούθησης θα ενισχύσουν τις αναγκαίες αλλαγές. Δεύτερο, θα πρέπει να ακολουθηθούν προσεκτικά οι γραμμές του προγράμματος. Να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομοθετικές προτάσεις μετά από εκθέσεις ιδίας πρωτοβουλίας. Τρίτον, η ιδέα είναι καλή, αλλά χρειάζεται να εξευρεθούν λύσεις εντός του χρονικού πλαισίου. Αναγκαία είναι επίσης και η διαφάνεια για τους διορισμούς εκπρές. Τέσσερα. Όσο μιλούμε για ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δημιουργούν απασχόληση, είναι σημαντικό να ενισχυθούν. Πέντε. Μελέτες αντικτύπου είναι αναγκαίες, αλλά μέσα σε κάποια χρονικά πλαίσια. Επίσης εδώ χρειάζεται διαφάνεια. Έξι κ. Καβαντά υποστηρίζει την πρόταση και για διαβουλεύσεις, δημόσιες διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενδιαφερομένων μερών. Τέλος, τελευταίο θέμα, οι αξιολογήσεις που κάνει το Συμβούλιο RSB θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και την αλληλεξάρτηση. Thank you for that. Ε, Jean... Ευχαριστώ πολύ. Jean Lambert απουσιάζει που κανονικώς ε, εκπροσωπεί του πράσινους. Κανείς δεν εκπροσωπεί την ομάδα η e EFTD. Επίσης, κανείς δεν εκπροσωπεί την Ευρώπη των Εθνών. Όμω η κυρία Ρέγνερ έχει ζητήσει το λόγο, η οποία τον λαμβάνει. Μάλιστα, έχω μία καταρχήν παρατήρηση για αυτό το λεγόμενο gold plating, αυτή την επιχρήσωση και τα, ε, τις προδιαγραφές. Αυτό το gold plating είναι απαράδεκτο. παραμορφώνει τα μέτρα Για μένα όμως έχει μεγάλη σημασία να γίνει διάκριση ανάμεσα σε αυτό το gold plating, αυτή την επιχρήσωση, κάτι το οποίο δεν έχει δηλαδή άμεση σχέση με το θέμα, και ελάχιστες, ελάχιστα πρότυπα, περί των οποίων και πρόκειται εδώ. Οι περισσότερες ρυθμίσεις για τις οποίες λαμβάνουμε νομοθετικές αποφάσεις εδώ για την προστασία των εργαζομένων, για τις συνθήκες εργασίας κλπ. Πολλά από τα οποία πολλά από τα όσα μάλλον αποφασίζουμε εδώ αποτελούν ελάχιστα πρότυπα. Όταν ένα κράτος και μια κυβέρνηση αποφασίζουν να εφαρμόσουν στο εθνικό δίκαιο μια οδηγία και να πούν ότι εμείς επιθυμούμε υψηλότερα πρότυπα, αυτό θα πρέπει να είναι δυνατόν πάντοτε να γίνεται στο εθνικό πλαίσιο. Κατ' επανάληψη είχαμε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που μας οδήγησαν στα όρια. Πρόκειται δηλαδή για ελάχιστα πρότυπα, είναι αυτά που θεσπίζονται δηλαδή, ή για ανώτατα πρότυπα. Έχει πραγματικά θεμελιώδη αξία. Χρειαζόμαστε ένα περιθώριο ως Ευρωπαίοι νομοθέτες. Πρέπει να διασαφίσουμε απόλυτα ότι βελτιωμένη νομοθεσία, better lawmaking, εδώ σημαίνει να βρεθούν βεβαίως απλοποιημένες λύσεις, αν είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρξουν κάποιες ε, αν υπάρχουν μάλλον ήδη κάποιες ρυθμίσεις, κάποιες λύσεις, να μην προσθέσουμε κι άλλες. Αλλά χρειάζεται να φροντίσουμε να μην ε, υπάρξει πολλαπλασιασμός των ρυθμίσεων. Είναι όμως αναγκαίο να υπάρχει περιθώριο υπέρ των εθνικών νομοθετών. Να είναι σαφές δηλαδή ότι αυτά που λέμε εδώ είναι ελάχιστα πρότυπα και βεβαίως το gold plating δεν έχει καμία σχέση με τα ελάχιστα πρότυπα. Η πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, έχουμε και εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που νομίζω ότι είστε εσείς κύριε ή κυρία Τζόνστον. Να μας πείτε όμως και το όνομά σας αφού λάβετε το λόγο. Λέγομαι Γιάννα Δεστούκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή της διαθεσμικής ε, συμφωνίας. Έχω δύο τεχνικά σχόλια. Αφενός επιθυμώ να αναφερθώ στην πολιτική συνάντηση, μάλλον στη συνάντηση πολιτικής καταγραφής που έγινε τον προηγούμενο Σεπτέμβριο και όπου συναντήθηκαν τα τρία θεσμικά όργανα και αναγνώρισαν την πρόοδο που έχει γίνει για την εφαρμογή του θεματολογίου της βελτιωμένης νομοθεσίας. Μετά υπάρχει και το ανακοινωθέν της 24 Οκτωβρίου όπου ανεβρίσκουμε την Annual Burden Survey σε ένα έγγραφο το οποίο επιγράφεται επισκόπηση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλοποίηση και βελτίωση του ρυθμιστικού, της ρυθμιστικής επιβάρυνσης. Άρα υπάρχουν αυτά, έχουν θεσπιστεί ήδη. Αυτά και μετά το υπαριθμόν 8, το διαθεσμικό μητρό ε, νομοθετικών πράξεων, το οποίο μάλιστα αναγνώρισαν τα τρία θεσμικά όργανα ότι πρόκειται για ένα υποδειγματικό εργαλείο διοργανικής συνεργασίας. Αυτά ήταν όλα που ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ. Thank you for that. Ε, η σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα για την εν λόγω έκθεση έχει ως εξής. Η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι η 29η πρώτου, το μεσημέρι ακριβώς. Έγκριση στην ΕΜΠΛ 21 με 22 Μαρτίου και μετά 27 Μαρτίου η έγκριση στην αρμόδια επί επιτροπή που δεν είμαστε εμείς. Μπορείτε θέλετε να πείτε εσείς κάτι κύριε Μακιντάιρ, αν θέλετε βεβαίως, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ναι. Ευχαριστώ όλες και όλους. Λέω στην Εύλη Ρέγνερ ότι συμφωνώ. Αν με είχε ακούσει για τα μεταλλαξιογόνα, θα είχε ακούσει να λέω ότι οι χώρες μέλη προχωρούν και παραπέρα. Εμείς δεν μπορούμε να τους πούμε όχι, μην προχωρήσετε περισσότερο. Προσπαθούμε να θεσπίσουμε τα καλύτερα δυνατά πρότυπα. Δεν αναφέρομαι όμως σε αυτό. Εγώ μιλώ για το gold plating εδώ που σημαίνει ότι προστίθεται και άλλα, πράγματα από πάνω τα οποία δεν έχουν ε, καμία θέση στα συγκεκριμένα πρότυπα και απλώς δυσφημούν την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Η Εύλην δεν επιθυμεί να επανέλθει καλώς. Μήπως άλλος κανείς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συμμετοχή σας στη συζήτηση που σημαίνει ότι προχωρούμε στο υπαρχόμενο 8 της ημερήσιας διάταξης που είναι η ακρόαση υποψηφίων για διορισμό εμπειρογνωμόνων στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Εκπαιδεύσεως. Είναι άραγε υποψήφοι εδώ. Είμαστε βέβαια και 10 λεπτά πιο πριν να περιμένουμε να προσέλθουν και οι τρεις υποψήφιες οι υποψήφοι. Βλέπω την Eddie Powers, τον Eddie Powers, τον Αλεχάνδρο Σέρκας. Και ο Ζαν francois Μετσιέ που δεν είναι εδώ. Μπορώ να παρακαλέσω λοιπόν την κυρία Μπάουερ να προσέλθει, αλλά παρόλα αυτά να περιμένουμε λίγα λεπτά ώστε να προλάβει να έρθει ο κύριος Σέρκας.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 Uh, Έχετε μείνει ελάχιστοι. Αυτό διευκολύνει τα πράγματα για την κυρία Μπάουερ και τον κύριο Σέρκας. Γνωρίζουν όμως πολύ καλά το σοβαρόν της συζήτησης αυτής, ανταλλαγή ε, απόψεων, με τους υποψηφίους ως ε, ε, εμπειρογνώμονες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Ίδρυμα για τις επαγγελματικές μαθητείες. Ε, ο κύριος Μεζιέρ δεν μπορούσε να είναι στην παρόν στη συνεδρίασή μας, όμως να δώσω το λόγο στους υποψηφίους που είναι παρόντες και παρούσες και στους λίγους βουλευτές που έχουν απομείνει στην αίθουσα Και επίσης γνωρίζουμε ότι παρίσταται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να δώσω το λόγο σε εσά, ε, κυρία Μπάουερ. Και να είστε βέβαιοι ότι σα παρακολουθεί ένα σωρό κόσμο που δεν είναι στην αίθουσα τώρα, αλλά βρίσκονται μπροστά στου υπολογιστέ του. Κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, συνάδελφοι. Όπως ξέρετε ήμουν μέλος αυτής της Επιτροπής 10 χρόνια. Και είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Όταν έφυγα από το Ευρωκοινοβούλιο, εξελέγηναν ανεξάρτητη εμπειρογνώμων για το Ίδρυμα αυτό. Εκτιμώ ιδιαίτερος το να μπορώ, την υπηρεσία αυτή μπορώ να σας προσφέρω και να σας εκπροσωπώ και να προσφέρω και την ε, όποια μου δουλειά στο οργανισμό αυτό, το ETF. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε για αυτόν τον οργανισμό είπα ότι παρόλο που βρίσκεται στα όρια των αρμοδιότητων αυτής της Επιτροπής στο ETF διότι επικεντρώνεται σε χώρες που δεν είναι κρατημέλη. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά σας. Τη δουλειά τους μάλλον. διότι έχουν πάρα πολλές γνώσεις και πολύτιμη εμπειρία για την απασχόληση από τη μια και τις πολιτικές ανάπτυξης από την άλλη. Βλέπω το ETF ως έναν οργανισμό που είναι ένα δυνατό εργαλείο για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας. Βλέπουμε τα προβλήματα με τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια στο μέλλον θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε αυτό το εργαλείο. Αυτό το τόσο κατάλληλο εργαλείο και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ε, λύσουμε αυτό το ζήτημα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις χώρες που δέχονται μεταναστευτικές ροές. Πανταχόφεν. Ο οργανισμός αυτός ε, εργάζεται υπό μεγάλη πίεση και ε, υπό το καθεστώς δημοσιονομικών περικοπών και μείωση του προσωπικού χρόνο το χρόνο. Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις τους είναι πολύ καλές και οι δραστηριότητές τους είναι και ενδιαφέρουσες και επικοδομητικές στις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής τους, παρά το γεγονός ότι το προγραμματισμός τους είναι ιδιαίτερα περιοριστικός. Έχουν εκατοντάδες αιτήματα, δηλαδή μέρα παραμέρα κάποιο αίτημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη μια καταλαβαίνω ότι πρόκειται για υπερβολικό φόρτο, Από την άλλη βλέπω ότι καμαρώνουν διότι συχνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει στην δική του την στήριξη, στην ε, βοήθεια λόγω της πολύ διαφορετικής κατάστασης που επικρατεί στα διάφορα κράτη. Θα ζητήσω λοιπόν την εμπιστοσύνη σας αύριο και βλέπω τη δουλειά μου ως μια προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ αυτής της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου και του ETF. Πραγματικά είναι πολύ καλή αποτίμησή μου προς τις επιδόσεις αυτού του οργανισμού. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ και τώρα ο λόγος στον κύριο Σέρκας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, βουλευτές ε, και λοιποί. Όπως είπε και η κυρία Μπάρ, θα ξεκινήσω και εγώ υπενθυμίζοντας ότι γνωρίζω πολύ καλά το Κοινοβούλιο. 15 χρόνια μακρά χρόνια από τη ζωή μου πέρασα εδώ, αν και μου φάνηκαν τότε πάρα πολύ σύντομα. Ε, θυμάμαι, ε, έχω πάρα πολύ ευχάριστες ε, αναμνήσεις και είμαι πολύ ευγνώμων για αυτά τα χρόνια. Όταν έλαβα αυτή την πρόσκληση από τους συντονιστές της Σοσιαλιστική ΟΜΑΔΑΣ για να συμμετέχω στην οργανισμό τωρινό Ανεξάρτητος εμπειρογνώμων. Ήμουν, έμεινα έκπληκτος αλλά είμαι και πάρα πολύ ευτυχής επειδή πλέον έχω πάρει σύνταξη, δεν φανταζόμουν πότε θα ξαναγυρίζα εδώ. Φανταστείτε την έκπληξή μου λοιπόν να επανέλθω στα παλαιό μου πάθος ε, και να ξαναβρω εδώ ε, στα έδρανα ανθρώπους με τους οποίους έχω μοιραστεί τόσο πολλά πράγματα κατά το παρελθόν. Και εγώ ε, είχα την πρόθεση να μην αναλάβω άλλο δημόσιο αξίωμα, αλλά ο οργανισμός, το Ίδρυμα του Τωρίνου ήταν αυτό που μου έδωσε το λόγο ε, γιατί είχα την, πάρει την απόφαση να αλλάξω σελίδα στη ζωή μου να παραβώ αυτή την ε, υπόσχεση. Γιατί έχει δύο ε, όψεις. Έχει το την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση αφενός αλλά και την ανεπτυξή συνεργασία ω αρμοδιότητε. Αυτό το ίδρυμα είναι πολύ προσφυλή θέματα για μας και για οικογενειακούς λόγους γιατί κατάγομαι από οικογένεια δασκάλων, παιδευτικών και να σας ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα θέματα της διαβίου μάθησης και εγώ που είμαι νομικός, θα δείτε βέβαια και τις λεπτομέρειες των βιογραφικών που έχω στείλει στην γραμματεία, αλλά έχω υπάρξει και εκπαιδευτικός, έχω διδάξει στο σχολείο και τώρα που πήρα σύνταξη ως βουλευτής ξαναγίνομαι πλέον εκπαιδευτικός και διδάσκω στο Πανεπιστήμιο στο Ζαμονέ, υπάρχει μια ενότητα Ζαμονέ στο Πανεπιστήμιο στη χώρα μου και αυτό κάνω. Και αυτό κάνουμε πολύ μεγαλύτερη σε ηλικία, ανακυκλωνόμαστε ε, και προσφέρουμε όπου μπορούμε τις υπηρεσίες μας. Ε, το Ίδρυμα λοιπόν ε, του Τωρίνου έχει μεγάλη σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και μου δίνει τη δυνατότητα να εργαστώ σε ένα τομέα πάρα πολύ προσφυλή για εμένα. Ξέρω πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση για τη ζωή ε, του ανθρώπου για τους λαούς. Ξέρω ότι το κοινωνικό συμβόλαιο που έκανε μεγάλη την Ευρώπη έχει ένα πολύ σημαντικό ε, κομμάτι που κανείς νομίζω δεν θέλει να αφήσει στην τύχη του. Μετά μιλάμε για το γύρας, ε, μιλάμε για την υγεία, λοιπά. Όμως έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, μια άλλη όψη. Τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν πλέον ε, τις ευκαιρίες για να προσφέρουν στην κοινωνία. Αυτό προσφέρει το Ίδρυμα, προσφέρει δεξιότητες ε, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται ε, με άλλους. Και θα ήταν αδικία να μην έχουν τις ίδιες δυνατότητες και ευκαιρίες. Υπάρχει μια κοινωνική αλλαγή, υπάρχει μια πολιτισμική αλλαγή και η συνεχής επιμόρφωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μελλοντικές προκλήσεις και για τις χώρες που βρίσκονται στον περίγυρό μας και που είναι και αντικείμενο του ε, Ιδρύματος του Τωρίνου. Η εκπαίδευση, κατάρτιση και το γνωρίζω πάλι από προσωπική εμπειρία είναι ίσως ε, η μόνη του ελπίδα, η μεγαλύτερη του ελπίδα τέλο πάντων για να καλύψουν το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των αναπτυσσόμενων ή πανάπτυκτων θα έλεγα χωρών και των δικών μα χωρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την εξωτερική τη διάσταση, την ε, συνεργασία και την ανάπτυξη ε, τα αντιμετωπίζει με πολύ καλό τρόπο και πραγματικά ε, θα νιώσω ιδιαίτερο ευτυχή αν μπορέσω κι εγώ εφόσον ψηφίσετε βέβαια να μπορέσω να βάλω το δικό μου λιθαράκι στο έργο που κάνει το Ίδρυμα για τις γειτονικέ μας χώρες. Αυτές είναι υποκειμενικές, είναι υποκειμενικοί μου λόγια. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ήμουν και στο τωρινό συντονιστή ε, τη Αλληλιστικής ομάδα. ξέρω το Ίδρυμα ε, και έχω διαβάσει και τη βιβλιογραφία του, τα συγγράμματά του, τα τελευταία αποτελέσματα των εξωτερικών εξολογήσεων, τα έχω μελετήσει. Νιώθω πάρα πολύ κοντά στο έργο του Ιδρύματος ε, και στα άτομα που εργάζονται εκεί, τα οποία φέρνουν σε πέρα μια αποστολή με στόχου αξιέπαινου κατ' εμέ. Γιατί στον Τωρίνο τι ξεκινά. Ξεκινά να υλοποιείται μια πραγματική δέσμευση. Δεν βασίζεται μόνο στη θεωρία αλλά και στην πράξη. Για μια καλύτερη Ευρώπη αλλά και καλύτερες γειτονικέ χώρες. Το Ίδρυμα στηρίζει πολύ ξεκάθαρα την εξωτερική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς που πρεσβεύουμε δεν θα μπορέσει να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια νησίδα ευημερία σε έναν ωκεανό εξαθλίωσης και άγνοιας. Το ίδρυμα τώρα και αποστολή του Τωρίνο είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Κάποιοι μπορεί να γίνουν μέλη της Ένωσης αλλά κάποιοι μπορεί να παραμείνουν γείτονε. και παρόλα ό,τι και αν συμβαίνει από τα δύο. Δεν θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα κλειό εξαθλίωσης και άγνοια αλλά ε, να δημιουργήσουμε γύρω μας ένα περιβάλλον με ανθρώπους που θα έχουν ελπίδα. Τι κάνουν οι Μαροκινοί που βλέπουν 16 χιλιόμετρα από τα σύνορά τους, ε, τα στενά το Γιβραλτάρ, ε, τι κάνουμε στην Ισπανία εμείς όταν εμείς μιλάμε για τα προβλήματα της ανεργίας, αλλά εκεί στο Μαρόκο ε, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι ξαφλιωμένοι που οι μόνοι λύση που βλέπουν είναι να μπουν σε μια σχεδία και να πνιγούν ε, προσπαθώντας να φτάσουν στην Ευρώπη. Νομίζω ότι με το ίδρυμα του Τωρίνου και την προσπάθειά του ε, ανακτούμε την αξιοπιστία μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε λοιπόν να στηρίξουμε τις μεγάλες ιδέες και στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να στηρίξουμε τις δυνατότητες αυτές των χωρών και εγώ πραγματικά είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένο αν μπορέσω, θα είμαι πολύ ικανοποιημένο αν μπορέσω να στηρίξω την εξωτερική διάσταση, την εξωτερική δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να τη δώσω την αξιοπιστία ε, και την νομοποίηση που ίσω ε, δεν έχει ακόμη. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική αξιολόγηση που είχε γίνει όταν ήμουν εγώ συντονιστή από το Ίδρυμα Δημοσίων Πολιτικών και Διαχείρισης για το Ίδρυμα του Τωρίνου. Διάβασα αυτή την αξιολόγηση και χαίρομαι γιατί δεν μπορούσαν να είναι πιο θετικά και ευνοϊκά τα σχόλια. Λέει ότι εξαιρετικά τα αποτελέσματα παρά το ευρύ ε, της ε, εντολής, είπε και η κυρία Μπάουερ, ότι έχουν να αντιμετωπίσουν στο Ίδρυμα πολύπλοκες καταστάσεις, δύσκολες, παρά την ευρύτατη εντολή και τους περιορισμένους πόρους, γιατί εκατομμύρια ε, είναι ο προπολογισμό του Ιδρύματο. Δεν φτάνει και για πολλά. Παρ' όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά άριστα. Θα ήθελα να στηρίξω λοιπόν το έργο που κάνει το Ίδρυμα και ιδίω ε, σε θέματα που είναι απόρρια και των αξιολογήσεων αυτών, ε, δηλαδή πού μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε. Υπάρχουν συστάσεις, τις έχω μελετήσει, που λένε ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η πληροφόρηση, η επικοινωνία και τα συστήματα δικτύωσης, τα δίκτυα. Το κάνουμε και εδώ, έχουν κάνει και άλλοι εκτελεστικοί οργανισμοί και άλλα ιδρύματα να μην περιοριζόμαστε στα του οίκου μας. Η αποστολή μας είναι πιο έξω, έξω από τους στίχους ε, των ε, θεσμικών οργάνων. Μην ομφαλοσκοπούμε ε, και ξεχνάμε τους άλλους. Υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν εκτός των τυχών της Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Θέλουμε να βελτιώσουμε λοιπόν τα εργολία, εργαλεία που μας συνδέουν, μας φέρνουν πιο κοντά στους πολίτες και εκεί θα εστιάσουμε. Επίσης υπάρχει κάτι πολύ ξεκάθαρο Στη διάρκεια της κρίσης όλοι οι εκτελεστικοί οργανισμοί και το Ίδρυμα προκειμένου ε, υπέφεραν από τη λιτότητα. Θα ήθελα λοιπόν να βοηθήσω σε σχέση και με το έργο του Κοινοβουλίου να βελτιωθούν ε, τα στοιχεία και η εικόνα αυτή. Επίσης θα ήθελα με ταπεινότητα μεν, αλλά και μεγάλο ενθουσιασμό να εργαστώ για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Εγκαλματικής Κατάρτισης, ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό ε, πιο αποδοτικό στη χρήση των πόρων του, να παγιώσει τη φήμη του, να μην βλέπει μόνο προς την Κομισιόν και τους υπαλλήλους της, αλλά τη φήμη του να την δημιουργεί, να την οικοδομεί εκτό. Στην κοινωνία δηλαδή τη ευρωπαϊκή. Ένωση. Είναι ένα πραγματικό κέντρο αναφοράς εξειδικευμένο στην ανέλυξη του ανθρώπου που επομένω θα μπορεί να ομιλεί με την ίδια δύναμη που το κάνει εντός και εκτό Ένωση. Οι παρεμβάσει του ιδρύματο ε, είναι διαρθρωτικού πολιτικού χαρακτήρα και νομίζω ότι η εμπειρία που έχω αποκτήσει εδώ στο Κοινοβούλιο θα με βοηθήσει να ε, δώσω τη δική σας φωνή να ακουστεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν μου δώσετε αύριο αυτήν την ε, ψήφο εμπιστοσύνη. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Σέρκαση. Κύριε Ρέγνερ, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Χαίρομαι πολύ που βλέπω και τους δυο σας εδώ. Νομίζω ότι Πραγματικά πρόκειται για θαυμάσιες υποψηφιότητες, απολύτως αξιόπιστες. Κυρίως γνωρίζω βέβαια τον Αλεχάνδρο Σέρκας και θα είμαι απολύτως ικανοποιημένη. Δεν ξέρω κανένα πρόσωπο που να έχει καλύτερο πολιτικό αισθητήριο, εμπειρία, ε, μεγάλη καρδιά αλλά και πείσμα για να προωθήσει τα θέματα αυτά. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που είχα την ευκαιρία να σας ακούσω και τους δυο σας εύχομαι καλή επιτυχία ήδη και ακόμη βέβαια κάτι που είναι σημαντικό ιδίως για μας εδώ τους ευρωβουλευτές ε, να είστε πάντοτε πείσμονες και να αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να κάνει κανείς κάθε δυνατή προσπάθεια ιδίως για τους οργανισμούς γνωρίζουμε ότι αποδίδουν εξαιρετικό έργο όμως καμιά φορά δεν είναι τόσο ορατό ε, γι' αυτό λέω σε αυτή την καθημερινή σας ζωή να ενοχλείτε ώστε να σημειώνουν τι κάνετε όλοι. Ε, χαίρομαι λοιπόν και πάλι που σας βλέπω και ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να με επιτρέψετε όμως να συνεχίσω στα Ισπανικά σαν ε, ε, να έχουμε κοινωνήσει πρώτη φορά μαζί με τον κύριο Σέρκας. Μπορεί και να μην το ψήφιζα ποτέ, δεν θα το σκεφτόμουν, αλλά είναι πολύ καλός μου φίλος και θα τον ε, ε ψηφίσω αύριο, όπως και οι άλλοι θα τον ψηφίσει αύριο, γιατί όλοι γνωρίζουμε τι δουλειά έχει κάνει εδώ πόσο σοβαρός ε, ε, το κύρος του, την ικανότητά του, ε, την εργατικότητά του. Αυτό που θέλω να πω εγώ και στους δύο είναι πρώτα απ' όλα ότι τους ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν να αναλάβουν αυτό το καθήκον. Και θέλω να τους πω και κάτι ακόμα σε σχέση και με τα όσα είπε η προλαλήσασα. Ναι, βεβαίως και πρέπει να γίνουν πολλά και πολλέ φορέ οι οργανισμοί κτλ. Όμως, υπάρχει και κάποια άγνοια σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο ως θεσμό και τη σχέση του με τα ε, θεσμικά ε, όργανα. Ε, το Eurofound, με το οποίο έχω εγώ, από το οποίο έχω εμπειρία, κάποιες φορές δεν υπάρχει γνώση επαρκής. Νομίζω ότι είναι ανεξάρτητα, δεν είναι αυτά και τα λοιπά. Και έτσι θα πρέπει να είναι. Δηλαδή, σας ζητώ να μην έχετε την αρχή να μην συνδέσετε άμεσα με το κοινοβούλιο. Καλό είναι το Ίδρυμα να αξιοποιείται και να λαμβάνετε περισσότερο υπόψη από το Κοινοβούλιο. να έχετε να προσφέρετε πραγματικά κάτι και να μην σας προσάψουν ποτέ τίποτε. Σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να λάβετε αυτή την ευθύνη και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Thank you. I'll give the floor to Madam Ευχαριστώ. Ο λόγος στην κυρία Μάκεντάιρ. Ευχαριστώ. Δεν είχα σκοπό να πάρω το λόγο, αλλά ήθελα να καλωσορίσω εδώ σήμερα τους πρώην συναδέλφους και να πω ότι είναι πολύ ευχάριστο να βλέπει κανείς ότι υπάρχει ζωή αφού πάψει κανείς να είναι ευρωβουλευτής. Χαίρομαι που έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μας και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω με τον κύριο Σέρκας. Ή τέλος πάντων συμφωνώ περισσότερο μαζί του σήμερα από τις προηγούμενες ευκαιρίες που συζητήσαμε. Πάντως, είναι πολύ καλό να γνωρίζω ότι οι δύο ψήφοι είναι εξίσου αξιόλογοι και ότι έχουν ε, προταθεί και οι δύο για τη θέση αυτή. Σας εύχομαι καλή τύχη. Thank you all and ε, we Ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σας αυτά. Ελπίζουμε λοιπόν να σας ξαναδούμε σε διαφορετικό πλαίσιο τα επόμενα χρόνια και ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Απολαύστε τα ε, αγαθά αυτά συναισθήματα απέναντί σας. Ε, έχοντας τώρα πει αυτά νομίζω ότι φτάσαμε και στο τέλος της ε, συναντήσεώς μας. Ευχαριστώ όλες και όλους που μείνατε έως τώρα. Και αύριο θα συνεχίσουμε και με ψηφοφορία. Αν και ορισμένοι από εμά θα προχωρήσουμε τώρα στον πέμπτο τριμερή διάλογο για την ε, απόσπαση εργαζομένων. Έχουμε ακόμα δηλαδή λίγες ώρες δουλειά. Θα σας ξαναδώ πολύ σύντομα. Ευχαριστώ για την συμμετοχή.